Good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί καλεσμένοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με τη δημόσια ακρόαση. Πρώτο σημείο της ημερήσης διάταξης η έγκρισή της. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις εγκρίνεται. Δεύτερο θέμα, έγκριση πρακτικών της συνεδρίας 18 και 19 Απριλίου του 2016. Και τρίτο, ανακοινώσεις Προέδρου. Τρεις Καταρχήν, δημόσια κρόση της Επιτροπής Αλίας για τη σημασία της αλίας ε, και κοινοτική και τοπική για γυναίκες τρίτων χωρών. Θα γίνει στις 15 Ιουνίου από 4 μέχρι 6.30 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών ε, έχουν προσκληθεί στη συνεδρίαση. Θα μας εκπροσωπήσει επισήμω ο αντιπρόεδρός μας, ο κύριος Ζωάου Πιμέντα Λόπες. Δεύτερη δημόσια κρόση, ή ε, μάλλον δημόσια συνάντηση, συνεδρίαση, Τη ομάδας εργασίας για την βία κατά των γυναικών. Θα γίνει μια τέτοια δημόσια συνεδρίαση τη Ομάδα Εργασία τη Επιτροπή ΦΑΜ με θέμα την βία κατά των γυναικών στι 21 Ιουνίου, 3 με 4.30 το απόγευμα, με θέμα την κύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. ο τίτλος της συνεδρίασης είναι «Προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, να κάνουμε την Ευρώπη ε, χώρο απαλλαγμένο από τη βία. Θα εκπροσωπηθούν το Συμβούλιο τη Ευρώπη, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, η Προεδρία και φυσικά οι συνεισηγητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα τη προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύμβαση αυτή. Θα σα μοιραστεί και στη ΦΑΜ και στη ΛΥΜΠΕ η, η ημερήσια διάταξη. Τώρα, το θέμα τη συνεκτίμηση τη διάσταση του φύλου στι πανεπιστημιακέ και ερευνητικέ οργανώσει θα γίνει μια υψηλού επίπεδου ε, διάλεξη με οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για Ισότητα των Φύλων στις 20 Οκτωβρίου του 2016. Σε αυτή τη συμμετέχουν 170 ηθήνοντες ε, ε, και αρμόδιοι για λήψη αποφάσεων, εμπειρογνώμονε, επαγγελματίε, αρμόδιοι για θέματα συνεκτίμηση διάσταση του φύλου στον ερευνητικό τομέα. Τα μέλη τη Επιτροπή μα προσκαλούνται συνεδρίαση και θα γίνει και εκδήλωση σε σχέση και με την τελευταία έκθεση κυρίας Βόζεμπερκ για τι γέλιε οροφέ που συναντούν οι γυναίκες ε, στη σταδιοδρομία του κυρίω στην επιστήμη και στα πανεπιστήμια. Και περνάμε στο κυρίως θέμα, το σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες της Ανατολικής ε, της ε, εταιρικής σχέσης, της ανατολικής σχέσης και άλλες γειτονικές χώρες. Στις 23 Νοεμβρίου του 2015 λάβαμε την έγκριση από το Προεδρείο για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης στα πλαίσια του πρώτου εξαμήνου του 2016 και θα αποτελέσει η ακρόαση αυτή ε, βάση για την προετοιμασία της δικής μας μη νομοθετικής ε, έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας για την οποία υποφαινόμενη είναι και η συγγήτρια. Και μάλιστα οι συντονιστέ αποφάσισαν στη συνεδρίαση τη 19η Απριλίου να προσκαλέσουμε την κυρία Μαριάννα Κατσάροβα επαμοιβή, ενώ οι υπόλοιποι ομιλητέ ήρθαν αφιλοκερδό. Θα έχουμε πολύ σημαντική ευκαιρία και χαιρόμαστε για αυτή τη δυνατότητα. Το κύριο θέμα είναι η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών ε, στις χώρες που καλύπτονται από τη χώρα Τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, που είναι χώρες ανατολική εταιρική σχέση, Μολδαβία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Αρμενία, Γεωργία και Αζερβαϊτζάν και οι χώρες της ε, Νότιας εταιρική Σχέσης, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, ε, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Ουκρανία, την Αλγερία, Λιβύη και Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων και σχέση με τις χώρες αυτές και να στηρίξει μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και του Μηχανισμού διάφορα ε, σχετικά σχέδια. Βέβαια, θα ασχοληθούμε με τα θέματα της οικονομικής χειραφέτησης, της βίας κατά των γυναικών, γιατί η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στις διάφορες χώρες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές επίσης είναι διαφορετικά. Μάλιστα, η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία θα πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή διαφοροποιημένη προσέγγιση στι γειτονικέ μα χώρε. Και περνάμε στην ακρόασή μα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εαυτό μου, μια και όπω σα είπα είμαι και η συγκίτρια αυτή τη έκθεση. Και θα περάσω τώρα στα γαλλικά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες ε, που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν εδώ την συνεδρίαση για τη συνεισφορά τους ε, στο θέμα των δικαιωμάτων των γυναίκων γυναικών ε, στις χώρες της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, και τις γειτονικέ χώρες. Όταν μιλάμε για τη γειτονία, για μένα είναι δύο οι λέξεις κλειδιά. σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να πάμε και πιο μακριά και να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή πορεία. Γιατί, Γιατί οι χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Είναι χώρες που έχουν μια σχέση εταιρική, βιώσιμη και αηφόρο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες από αυτές ε, ε, δεν είναι μόνο μέρος της εταιρική ανατολικής σχέσης, αλλά έχουν μπει και στην ευρωπαϊκή πορεία. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από κοινέ αξίες, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των ανθρώπων και τη δημοκρατία. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν ένα κοινό σημείο των χωρών αυτών είναι ότι είναι χώρες σε μετάβαση ή ότι θέλουν να κάνουν βαθιές μεταρρυθμίσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Γειτονίας είναι σε μια τριπλή μετάβαση, πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογειακής ε, Γειτονίας είναι λίγο πιο ε, ομογενοποιημένες ως προς το πολιτικό του σύστημα και το κοινωνικό σύστημα. Θα μπω σύντομα τώρα σε μία δικαιολόγηση σχετικά με την κάλυψη της έκθεσης. Στο θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών και της συμμετοχής τους ε, ε, βλέπουμε ότι η κατάσταση και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές ε, στις διάφορες πολιτικές. Παρόλα αυτά υπάρχει μια κοινή μέθοδος και ένας κοινό στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία μιας σταθερής και σίγουρης γειτονίας και κατά συνέπεια ε, δημοκρατική που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των γυναικών. Γι' αυτό και η συγγήτρια, δεδομένου και του δεύτερου σημείου ε, του τίτλου, ε, Προσπάθησα στη σύνταξη της έκθεσης ε, να συμπεριλάβω και τις χώρες ε, της νότιας πολιτικής γειτονίας. Αυτή η πολιτική είναι υπό αναθεώρηση και υπάρχει λοιπόν μια σημαντική ευκαιρία να βάλουμε τα δικαιώματα, τη χειραφέτηση και τη συμμετοχή των γυναικών στις προτεραιότητες. Προσπάθησα λοιπόν από τη μία να επικεντρωθώ στην ανατολική εταιρική σχέση, αλλά μην εξαιρέσω και τις νότιες χώρες ε, που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, αλλά ούτε και τη θέση των γυναικών σε αυτή την πολιτική. Η συμβολή των εμπειρογνώμων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης θα μας επιτρέψει να προτάξουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των διαφορών πολιτικών γειτονίας. Όμως όλα αυτά δεν θα μας εμποδίσουν τελικά να έχουμε μία ε, έκθεση στο νότιο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας. Ε, οι χώρες που δεν είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής γειτονίας, όπως είναι οι Βαλκανικές χώρες, η Τουρκία και η Ρωσία, αντιμετωπίζονται μέσα στα πλαίσια των διμερών σχέσεων και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, άλλα μέσα λοιπόν. Επίσης, ε, προσπάθησα να δώσω έμφαση στη σημασία του θέματος. Για όσους είναι εδώ σε αυτή την αίθουσα, είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε λοιπόν όμως να το επαναλαμβάνουμε, ότι ο σεβασμός των, των δικαιωμάτων των γυναικών στις χώρες της γειτονίας ε, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, είναι μια κοινή αξία, μια κοινή φιλοδοξία και ε, θέλουμε ε, με αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε και την γειτονία η οποία θα είναι δημοκρατική και σταθερή. Τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες αυτές πρέπει να γίνονται σεβαστά de και de facto για να μπορεί η συμμετοχή τους ε, στην κοινωνική και οικονομική ζωή να είναι εγγυημένη. Η σταθερή πολιτική γειτονία είναι μια πολιτική που οδηγεί στην, στον πλούτο και την συμμετοχή των γυναικών. Θα τελειώσω την εισαγωγή μου με κάποιες ερωτήσεις για τους εμπεριγνώμενες και την Επιτροπή. Όταν ξεκινάμε να συντάσσουμε μία έκθεση, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το θέμα των δεδομένων και των αριθμών όσο προς τον σεβασμό των, των δικαιωμάτων των γυναικών, για τη... ως προς τη βία, τη συμμετοχή των γυναικών τα πολιτικά, περιφερειακά και τοπικά θεσμικά όργανα, όπως και η πρόσβασή τους ε, στη δικαιοσύνη. Ποια είναι τα δεδομένα. Αυτά θα θέλαμε οι εμπειρογνώμονες να μας δείξουν ε, για να μπορέσει η έκθεσή μας να αποτελέσει μια βάση που θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στην ε, προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Επίσης ενδιαφερόμαστε για τις βασικές προκλήσεις σε αυτές τις περιοχές. Όταν όμως μιλάω για προκλήσεις, ε, να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει ακόμα είναι και η δυνατότητα να δώσουμε και απαντήσεις σε αυτές, που θα είναι επαρκείς και θερεαλιστικέ. Ε, θα μπορούσαν οι εμπειρογνώμονες ξεκάθαρα να μας ε, δώσουν κάποια ένδειξη σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Τι είναι το πιο επίγον που πρέπει να γίνει και τι θα γίνει εν ευθέτω το χρόνο. Ποιοι είναι όλοι οι παράγοντες αυτοί, οι πολλαπλοί παράγοντες που θα μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Για την ε, ανατολική εταιρική σχέση επίσης υπάρχει το θέμα της ε, κληρονομιάς της κομμουνιστικής εποχής, η οποία, το οποίο βρίσκεται, η οποία βρίσκεται ε, στους θεσμούς υπάρχουν στερεότυπα τα οποία παραμένουν και επηρεάζουν και τα δικαιώματα των γυναικών. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που το εξηγούν αυτό. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τις μεσογειακές χώρες. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ε, θέληση για μεταρρύθμιση της πολιτικής ηγεσίας, αλλά είναι συντηρητικοί η ε, λαοί ε, στο Μαρόκο, στην Τινησία κτλ. Ποια είναι λοιπόν τα μέσα που η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονιά θα μπορούσε να κινητοποιήσει για να μπορέσουν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές να γίνουν με τη μέθοδο bottom-up, από κάτω προς τα πάνω, να μην είναι μόνο top-down, από την ηγεσία προς τα κάτω. Θα ήθελα επίσης ε, να δώσω έμφαση και στα εργαλεία και το πλαίσιο εργασίας που είναι πιο αποτελεσματικό για μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική γειτονία. Να είναι η έκθεση ένα βήμα μπροστά σε αυτό το θέμα. Και όταν μιλάμε για έκθεση, ε, μιλάμε και για βέλτιστες πρακτικές, άρα η ιδέα είναι να προωθήσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών ε, της ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης. Θα θέλαμε οι εμπειρογνώμονες να μας δώσουν παραδείγματα από τέτοιες πρακτικές, αλλά για να μπορέσει κυρίως να γίνει αυτή η ανταλλαγή θα πρέπει και εμείς ε, να σας ακούσουμε και να ε, δώσουμε ένα βήμα παραπέρα για να προασπιστούμε ε, τα αιτήματα των γυναικών. Αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν με το που ξεκίνησα την έκθεση. Ε, τώρα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψε, να δώσουμε απαντήσεις και θα ήθελα ε, εκ των προτέρων για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Είμαστε εδώ, ανυπομονούμε να ακούσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, σας, ε, τις απόψεις, την κριτική σας. Και χωρίς να μακρηγορώ άλλο, θα δώσω το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Ματεριάνα Κατσάραβα, που είναι ιδρύτρια και πρόεδρο του Reach All Women του uh, UK uh, and Society for Justice Foundation της Βουλγαρίας, uh, ιδρύματος δηλαδή για την κοινωνία και τη δικαιοσύνη. Να σας ευχαριστήσω γιατί εδώ και χρόνια έχετε εμπλακεί στον αγώνα κατά της βίας των γυναικών, προασπίζεστε τα δικαιώματα των γυναικών. Σας δίνω λοιπόν το λόγο και με ανυπομονησία θα ακούσουμε το μήνυμά σας. Ε, Thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάμπριελ, ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και για τις ερωτήσεις που μας θέσατε ως εμπειρογνώμονες. Ελπίζω να μπορέσουμε να απαντήσουμε και μάλιστα να δώσουμε απαντήσεις μεστές νοήματος. Σήμερα βέβαια δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά είμαι βεβαία ότι οι συνάδελφοι θα έχουν ε, κάθε καλή διάθεση να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας κατά τη σύνταξη της έκθεσης, σε εσά και τους συναδέλφους σας. Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω την ε, πρόεδρο, την κυρία Γκαρσία Πέρες, ε, ίσως να μην είναι εδώ σήμερα, για την ευγενική της πρόσκληση προς εμάς, τους εμπειρογνώμονες, αυτή την ακρόαση και ευχαρίστως να σε βοηθήσουμε, Μαρίγια, ε, γιατί ηγείσαι του αγώνος ε, στην Βουλγαρία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να πετύχουμε ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες στη χώρα μας. Ευχαριστώ και όλους σας, τα μέλη αυτής της Επιτροπής, για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και της Νότιας Γειτονίας. Διότι θεωρώ ότι η στιγμή είναι κρίσιμη. Πρέπει να ασχοληθούμε ακριβώς τώρα με αυτά τα προβλήματα. Να επικεντρωθώ σήμερα σε δύο ζητήματα από όλο το θεματολόγιο των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ανατολική και Νότια Γειτονία Δύο ζητήματα που συχνά τα παραβλέπουν οι πολιτικοί υφήνοντες στις συζητήσεις και τις αποφάσεις τους. Ένα, ε, τα βασικά αριθμητικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα βέβαια. Θα ήταν καλό να τα είχαμε, γιατί θα ήταν ένα καλό σημείο αφετηρίας για περαιτέρω έρευνα για τα θέματα αυτά. Πρώτο θέμα είναι ο ρόλος των γυναικών στην ε, ε, πάυση των εχθροπραξιών ή συγκρούσεων και στην οικοδόμηση συνθήκων ειρήνης και μετά είναι τα δικαιώματα των ακτιβιστριών για θέματα ειρήνης. Επίσης η έκτακτη προστασία που μπορεί να απαιτείται για αυτές και η παρακολούθησή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, ποιότητα στα δικαιώματα των γυναικών στην ευρωπαϊκή γειτονία. Είναι ουσιαστική σημασία για την ίδια την ειρήνη και την ασφάλεια για όλου στην Ευρώπη. Διότι η πολιτική ασφάλεια δεν είναι θέμα απλώ διοντολογικό ή ένα ηθικό δίλημα ή ένα θέμα τη επίτευξη πλήρου δικαιοσύνη. Η ισότητα των γυναικών είναι ζωτικό συμφέρον κάθε έθνου και του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Η ε, ισότητα η μη ισότητα, μάλλον η ανισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών και η διακριτική του μεταχείριση είναι απειλή για την ευστάθεια κάθε κράτου και για το συνολικό δρόμημα ασφαλεία του. Μίσος, βία και οργή είναι αυτό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν οι άντρε τους ε, πολεμούν. Πολλέ φορές είναι εκείνε που μαζεύουν τα σπασμένα και φροντίζουν ε, να ε, συνδέσουν τους δεσμούς της κοινωνίας τους. Ε, δικηγόροι, δικηγόροι, νοσοκόμες, κοινωνικές λειτουργοί, γυναίκες που εργάζονται πολλές φορές σκληρά με τα μηνύματά τους να περνάνε σαν μήνυμα σε μπουκάλι διότι ε, προσπαθούν να στηρίξουν τους άντρες και τα παιδιά τους. Μετά το δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας τη δεκαετία του 90, που δεν είναι ακριβώς η ανατολική μας γειτονία, είναι το ανατολικό μέρος της γειτονίας μας, εκεί συνάντησα τουλάχιστον 2.000 γυναίκες που βιάστηκαν από στρατιώτες. Και είδα πόσο νοπός ήταν ο πόνος τους, η οδύνη τους από τη βία που έζησαν στα χέρια αλλοδαπών στρατιωτών. Πόσο ντροπή και απελπισία αισθάνονταν, πόσο μοναξιά ταυτόχρονα πραγματικά έμεινα άναυδη με τη βούληση αυτών των γυναικών να ζήσουν, να επιβιώσουν και να εκφράσουν στον έξω κόσμο τον αποτρεπιασμό τους για τον πόλεμο. Να πούν τη δική τους ιστορία και να αποδώσουν δικαιοσύνη, να φέρουν την ειρήνη. Από το 2006 υπάρχει μια οργάνωση στην οποία βοήθησα στην ίδρυσή της, Regional Women in War, ή τέλο πάντων Raw in War ε, για την προστασία των γυναικών αυτών και την ψυχολογική του στήριξη. Γιατί συζητάμε το θέμα αυτό σήμερα. Διότι ομοία αλήθεια είναι ότι η ιστορία διεθνή κοινότητα δεν κατάφερε να ε, οικοδομήσει ειρήνη και ασφάλεια διαρκεία. Πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο πάνω από τι μισέ ειρηνευτικέ συμφωνίε στον κόσμο εντό πενταετία δεν οδήγησαν στα αποτελέσματά του. Τουλάχιστον 12 ένοπλε συγκρούσει βρίσκονται σε εξέλιξη στον κόσμο χωρί να μετράμε τι παγωμένε ή τι ε, σε κρεμότητα. Εδώ μόνο μία χώρα της Ανατολικής Μακεδονίας η Λευκορωσία δεν έχει αντιμετωπίσει ενόπλη σύγκρουση τα τελευταία χρόνια με τη μια την άλλη μορφή. ενεργέ εχθροπραξίε όπω στην ε, Ουκρανία, στα πρόθυρα ε, ανοιχτή σύραξη στον Αγκόργονο Καραμπάχ, με συγκρούσει μεταξύ Αρμενία και Αζερβαϊτζάν πρώτων θυρών, ε, ο αντίκτυπο του πολέμου στη Γεωργία και το τι συνέβη με τι συνέπειε του πολέμου στην Αμπχαζία και την Νότια ή την τη δημοκρατία της Μολδαβίας ε, και τον αντίκτυπο του πολέμου, βλέπουμε ότι έχουμε 700 χρόνια καθυστέρηση στο παγκόσμιο προπολογισμό του ΟΗΕ με τις στρατιωτικές δαπάνες ή 2.900 χρόνια του προπολογισμού του ΟΗΕ για τα θέματα των γυναικών. Και πάλι οι γυναίκες αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και από του ε, πολιτικού θεσμού που τι αναλαμβάνουν. Πραγματικά δεν πάβει να με εκπλήσει ότι αυτοί που έχουν συμμετάσχει στι ένοπλε εχθροπραξίε, που έχουν ε, αφαιρέσει τη ζωή ε, αμάχων ή με του αξιωματικού του έχουν σχεδιάσει τον επόμενο πόλεμο ή σύγκρουση, αυτοί είναι που κρατούν εχμάλωτο τι γυναίκε. 80% των θυμάτων και των προσφύγων πολέμου ή συγκρούσεων. Τις κρατάνε μακριά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπου φτιάχνεται, πλάθεται η συγκρουσεων τι κρατανε μακρια απο το Είναι παράλογο. Πού είναι ο ρόλο ε, των γυναικών στο τραπέζι αυτό που συζητιέται η ειρήνη. Είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε πολλά στοιχεία στα χέρια μα που δείχνουν ότι οι γυναίκε ανά τον κόσμο έχουν συμβάλει στην δημιουργία και διατήρηση τη ειρήνη. Ενώ η συμμετοχή του οδηγεί σε διαρκέστερα και βιωσιμότερα αποτελέσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό, όταν οι γυναίκε εμπλέκονται σε ειρηνευτικέ διαδικασίε, φέρνουν στο τραπέζι των συζητήσεων τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την συμφιλίωση και την ανακοδόμηση της οικονομίας ή βασικά στοιχεία, αλλά πολύ κρίσιμα, όπως την ε, υγιεινή, την επιστηστική ασφάλεια και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι το πρώτο στοιχείο που είπε ο Λιβεριανός πρόεδρος ε, Τζόνσον όταν ξαναπήρε την εξουσία ήταν ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί το αποχετευτικό σύστημα και να υπάρχει τρεχόμενο νερό στα νοικοκυριά στη Λιβερία. Τώρα πείτε μου, πόσοι ε, άρενες πρόεδρες ε, χώρες μετά από πόλεμο θα σκέφτονταν ως πρώτη προτεραιότητα αυτό. Και παρόλα αυτά οι γυναίκες το 2012 σε μια σχετική μελέτη βρέθηκε ότι στις 12 μεγάλες ελληνικές διαδικασίες από το 1992 μόνο σε 4% των υπογραφών που βρέθηκαν σε αυτές τις συμφωνίες ήταν γυναικείες. 2,4% των βασικών διαιτητών ε, ήταν γυναίκες, 3,7% των μαρτύρων ή παρατηρητών στις ελληνικές διαδικασίες ήταν ήταν γυναίκες, 9% των ε, ομάδων των διαπραγματευτών είχαν μέλη γυναίκε, οπότε προφανώ υπάρχει πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν αλλάζει τίποτα στι χώρε τη Ανατολική Γειτονία προφανώ. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκε δεν έχουν συμμετάσχει στις ιδιωτικέ διαδικασίες του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το 2012 τέσσερις γυναίκες εκπροσωπούσαν την αντιπροσωπεία τη γεωργία στι συνομιλίε τη Γενέβη από 10 συμμετέχοντε. Ε, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικείας συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητε. Σήμερα μόνο δύο έχουν απομείνει. Ε, όταν οι γυναίκε δεν συμμετέχουν, ε, όπω στη διαδικασία του Μίνσκ για την ένοπλη σύραξη στα ανατολικά τη Ουκρανία, με την εξαίρεση της κυρίας Μέρκελ βεβαίως στην επίσημη ιδιότητά της, βλέπουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών είναι αναγκαία στην ειρηνευτική διαδικασία. Οι γυναίκες επίσης απουσιάζουν από την ειρηνευτική διαδικασία στην ε, συνομιλίες για την ε, υπερνηστερία στη Μολδαβία. Επίσης οι γυναίκες απουσιάζουν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Συρία ε, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών. Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια πίεση από ομάδες γυναικών, το Μάρτιο του 2016 ανακοινώθηκε ότι οι 12 γυναίκες από την κοινωνία των πληκτών θα επιτραπεί να παρέστανται σε αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως μέρος ενός συμβουλευτικού μόνον σώματος. Αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα βέβαια, αλλά οι γυναίκες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μόνο στα περιθώρια των επίσημων συνομιλιών για την ειρήνη στη Συρία. Ε, Κυρίε και κύριοι, στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση και πάλι στα ανατολικά τη Ουκρανία. Δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ενημέρωση πλέον, αλλά πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εχμαλωτοί ε, στι περιοχέ του Λουγκάνσκ στα ανατολικά της Ουκρανίας με παραβιάσεις των θεμελιδών τους δικαιωμάτων ενώ υποφέρουν από διακρα... διακριτική μεταχείριση με ε, βομβαρδισμούς ε, με ε, αφαίρεση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, τη βασική επισητιστική ασφάλεια και τα βασικά τους δικαιώματα, καθώς και τις απειλές βασανιστήριων, απαγωγών, την απουσία ελεύθερης κυκλοφορίας. Μόλις επέστρεψα από την Ουκρανία, όπου βρισκόμουν τα τελευταία δύο χρόνια, όπου ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας στο Ντονέτσκ, στο Λουγκάντ, στο Γιέτνο Πετρόφσκ και και στη Μαριούπολη ε, επί δύο χρόνια του αρμόδιου φορέα του ΟΗΕ. Είδαμε τι έχουν υποστεί εκεί γυναίκε και κορίτσια, αλλά δυστυχώ λόγω του φόβου αντιπίνων οι γυναίκε δεν καταγγέλουν τον βιασμό. Η διακίνηση ανθρώπων, το εμπόριο ανθρώπων στην Ουκρανία επίση είναι ενεργό. Εκατομμύρια γυναίκε, άντρε και παιδιά γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτοι στην ε, εμπορία ανθρώπων. Όμω δεν υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα, ούτε έρευνε για το σχετικό φαινόμενο, ούτε προγράμματα και σχέδια για να στηριχθούν τα θύματα ε, η ένοπλη σύραξη στην Ουκρανία οδήγησε στην αύξηση τη ανδροκογενειακή βία, ε, τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην υπόλοιπη χώρα, λόγω τη αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση στην κοινωνία και του αριθμού όπλων και από τι δύο πλευρέ τη οπλοκατοχή δηλαδή. Βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλε τι ενόπλε σειράξει στον κόσμο και συμβαίνει και τώρα στην Ουκρανία. Ε, οι πρώην μαχητέ που είναι τραυματισμένοι, ε, τα αντίπεινα του τα εκφράζουν στην ε, κοινωνία με πρώτα θύματα και στόχο την οικογένεια και την ε, κοντινή τους, το κοντινό του περιβάλλον. Υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα όμω στο κατόφλι των γυναικών. Αυτό ο πόλεμο του Ισλαμιστικού κράτου κατά των γυναικών και κοριτσιών στο Μοσούλη, στο Ιράκ, πριν από μία εβδομάδα, 12 γυναίκε και κορίτσια ε, ε, κάηκαν στην πειρά σε σιδερένια κλουβιά γιατί αρνήθηκαν να είναι σεξουαλικέ σλάβε των μαχητών του Άιζη. Και 3.000 γυναίκε και κορίτσια στο βόρειο Ιράκ κρατούνται εχμάλωτε ε, στου σκλάβε του 6 για του μαχητέ ε, του Ισλαμικού κράτου. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό και στι διαπραγματεύσει να περιληφθεί το θέμα τη απελευθέρωσή του και τη ε, ψυχολογική του στήριξη για να μπορέσουν να αναρρώσουν. Σε γενικέ γραμμές, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι στις χώρε της Ανατολική Γειτονία, οι γυναίκε απουσιάζουν από τις ε, επίσημες θέσει εξουσία και λήψη αποφάσεων. Οι καλύτεροι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τα θέματα ισότητα των φύλων, ιδίω κατά των γυναικών, κατά την άποψή μου, είναι οι ίδιε οι γυναίκε σε πολιτικέ θέσει, σε θέσει πολιτική εξουσία. Ωστόσο, στι χώρε Ανατολική Γειτονία, λίγε είναι οι γυναίκε που έχουν πολιτική εξουσία. Έχουν αγωνιστεί τόσο πολύ για να φτάσουν ω εκεί, που τελικά το τελευταίο που θέλουν να κάνουν είναι να βγουν στην κοινή γνώμη και να μιλήσουν για θέματα που δεν είναι δημοφιλή. Όπω η βία κατά των γυναικών ή η ισότητα των φίλων. Ε, δεν θέλουν τη σφραγίδα των φεμινιστών από τους άντρες συναδέλφους τους ή από την κοινή γνώμη του. Να τις αποκαλέσουν φεμινίστριες είναι ένας όρος ε, μειωτικός στην Ανατολική Ευρώπη. Σημαίνει στα καλύτερη περίπτωση ότι είσαι ανεπιθύμητη και άσχημη και... Ε, ότι δεν έχεις αξία. Το ίδιο όμω θα έπρεπε να ισχύει και για έναν άντρα. Όσε γυναίκε έχουν καταλάβει θέσει εξουσία και λαμβάνουν αποφάσει στι χώρε τη Ανατολική Γειτονία, πρέπει διαρκώ να θυμούνται ότι έχουν έναν μοναδικό και αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσουν στην αλλαγή τη νομοθεσία και τη πολιτική για να βελτιώσουν τι συνθήκε ζωή των κοριτσιών και των γυναικών στη χώρα του. Πρέπει να υψώσουν τη φωνή του. Πρέπει να εκφραστούν δημοσίω και να στηριχθούν και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το κοινοβούλιο όταν είναι τόσο τολμηρέ στη δική του χώρα. Το θέμα τη ισότητα των γυναικών έχει αναποτεθεί στα χέρια τη κοινωνία των πολιτών κατά μεγάλο μέρο και τη ομάδα των γυναικών. Όμω αγωνίζονται για κονδύλια και πολλέ φορέ ε, επιβιώνουν με δυσκολία, μένοντα στο περιθώριο των δημόσιων και επίσημων συζητήσεων ή διαπραγματεύσεων. Η εχθρότητα κατά των γυναικών για την ανάληψη θέσεων εξουσία από αυτέ δεν μα εκκλείσει και δεν είναι, δεν είναι περίεργο που και στι ε, συνομιλίε για την ειρήνη οι γυναίκε δεν είναι πρόσδεκτε ε, όταν ε, μιλούν για τι ένοπλε συγκρούσει σε αυτή την περιοχή. Τι μπορεί περισσότερο να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν Πρώτον, η αλλαγή πρέπει να αρχίσει στι ίδιε τι χώρε μα. Από τι ε, εννέα ειδικού απεσταλμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί από του οποίου ε, συμμετέχουν στι ε, διεθνεί ειρηνευτικέ συνομιλίε και στι χώρε τη Ανατολική Γειτονία, ξέρετε πόσοι από αυτού του δέκα είναι γυναίκε. Καμία θα μπορούσε καλής να πει ότι η θέση της είπα της εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα χέρια μιας γυναίκας. Αυτό βέβαια δεν μας καλύπτει, διότι μιλάμε για γυναίκες που συμμετέχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χαράξει το δρόμο και να σταθεί ως παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Ως προς τις διαδικασίες ε, διορισμού, πρόσληψης, πρέπει να προσθέσονται τέτοιες θέσεις εργασίας και να είναι και πιο βιώσιμες. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα από γυναίκες υψηλών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι υποψήφιες για τέτοιου είδους θέσεις. Αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Επίσης, ε, προτείνεται η συμμετοχή ειδικών δικτών για τις γυναίκες στην εξουσία. Πόσες γυναίκες συμμετέχουν στις επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες. Υπάρχουν δύο βασικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τι γυναίκε τη ενόπλε σειράξη και τι γυναίκε τη ειρηνευτικές συνομιλίες από το 2006 και 2012. Έχουν υλοποιηθεί πλήρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ω προ τι χώρε τη Ανατολική Γειτονία. Για παράδειγμα, το ψήφισμα Δευτέρα Φεβρουαρίου 2016 καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τι ειρηνευτικέ συνομιλίε, ώστε να συμμετέχουν σε αυτέ και οι γυναίκε στι ομάδε των διεθνών διαπραγματευτών και σε ηγετικέ θέσει. Ζητά να επιτελεστεί πρόοδο στην μόνιμη συμμετοχή γυναικών ε, ε, ηγετιδών, εκπροσώπου από τι ε, τοπικέ ομάδε γυναικών και διαπραγματεύτριε στι διαδικασίε για την ειρήνη. Βεβαίω πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια του Κοινοβουλίου στη συμμετοχή των γυναικών στι ειρηνευτικέ συνομιλίε, να εξαρτάται να είναι ένας όρος και μια προϋπόθεση για όλα τα κράτη, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας. Το ίδιο ψήφισμα ε, συνιστά τη δημιουργία ειδική εκπροσώπου για τις γυναίκες της ε, ειρηνευτικές συνομιλίες στα πλαίσια της ΕΕ ώστε να είναι σταθερή η διάσταση της ισότητας των φύλων και να υπάρχει και συνεννόηση με τους ομολόγους των ΟΗΕ. Ε, επίσης συνιστά αυτό να ισχύει σε όλες τις ομάδες κρούσης και ε, γενικής διευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και όλα αυτά να αναφέρονται στην ειδική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρχει συνοχή και συνέπεια και επίσης συστηματική και συνολική υλοποίηση όλη τη στρατηγική που θα πρέπει να ε, αναλυφθεί και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικού συντονισμού. Θα μπορούσε να ενισχυθεί με την όθηση πραγματικά να διοριστεί ε, μια ειδική εκπρόσωπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη θέση ελπίζουμε να την κατέχει η γυναίκα βέβαια. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το να υπάρχουν ε, φορεί γυναικών που να συμμετέχουν στι ειρηνευτικέ συνομιλίε δεν σημαίνει ότι τα θέματα των γυναικών και η προοπτική των γυναικών θα συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία αναγκαστικά. Οι εκπαιδευμένε γυναίκε από την κοινωνία των πολιτών, οι πολιτικοί και οι βουλευτίνε από την Ανατολική γειτονία στι ειρηνευτικέ συνομιλίε και ε, τη Ανατολική και τη Νότια γειτονία με δεξιότητες για διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις που να είναι εκπαιδευμένες και προετοιμασμένες πώς να διατυπώνουν, να διαπραγματεύονται και να ε, προβάλλουν τα θέματα ισότητας των φύλων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και για τη συμπερίληψή του σε συμφωνίε για την ειρήνη είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι οι μελέτες δείχνουν ότι το ψήφισμα του ΙΕ 1325 από το Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν πραγματικά ε, ένα σημαντικό ε, εφαλτήριο για να αρχίσουν να συμμετέχουν οι γυναίκες σε τέτοιες ειρηνευτικές διαδικασίες όμως στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Μόνον στη Γεωργία το 2011 η Βουλή ενέκρινε για το 2012 έως 2015 ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης για τη γυναίκα στην ειρήνη και την ασφάλεια και ως προς την υλοποίηση του ψηφίσματος του ΙΕ 1325. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει όλες οι χώρες της Ανατολικής Ιδονίας να εγκρίνουν ένα εθνικό πρόγραμμα για το ψήφισμα του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΑ 1325, δημιουργώντας τον ανάλογο μηχανισμό για την παρακολούθηση της υλοποίησης των διτάξεών του. Τρίτον, να εργαστούμε με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους φορείς του ΙΕ, ώστε οι γυναίκες και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προσπαθειών ανακούφισης έκτακτων αναγκών, με τον σχεδιασμό της ανοικοδόμησης, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, αλλά κυρίως στη φάση μετά τη σύγκρουση πρέπει να αντιμετωπιστεί η ατιμορρησία για την εμπορία ανθρώπων, για το τι γίνεται μετά τις εχθροπραξίες, για το να μην ε, υποφέρουν κι άλλο τα θύματα γυναίκες και κορίτσια και κυρίως να μην μένουν αόρατες ε, στην περίπτωση χωρών που έχουν περάσει από ένοπλες συγκρούσεις. Μηχανισμοί για τον εντομισμό των θυμάτων και για την παροχή ε, κατάλληλη προστασία είναι επίση κάτι απαραίτητο. Η οικονομική στήριξη των γυναικών σε διάφορε κοινότητε που βγαίνουν από συνθήκε πολέμου και συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει σε ευμάρεια ολόκληρο έθνο με την καταπολέμηση τη εμπορία και τη εκμετάλλευση. Και τέλο, πρέπει να προσφερθεί κατάλληλη και στοχευμένη χρηματοδότηση για τι ομάδε γυναικών και τι ε, αυτόρμητε ε, ε, αυτό με οργανωμένε ομάδε σε χώρε ε, συγκρούσεων ή μετά από εχθροπραξίε στι ε, χώρε τη Ανατολική και Γειτονία. Μηχανισμοί χρηματοδότησης που να είναι ευέλικτοι και εύχρηστοι με στόχευση στα γυναικεία μέλη των κοινοτήτων είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Το να ακούσουμε τις γυναίκες από την κοινωνία των πολιτών και τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, γιατί πρέπει να γίνει στις χώρες μετά από συγκρούσεις ή κατά τέτοια των συγκρούσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό και με επίσημη επικοινωνία μαζί τους για την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη των ενοπλών συγκρούσεων. Η και η κατάρτιση εκθέσεων για τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών. Οι για την ανάδυση ένοπλων συγκρούσεων, η στήριξη με χρηματοδότηση και μηχανισμό προστασία για τι γυναίκε που είναι ακτιβίστρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αντιμετωπίζουν απειλέ κατά τη ζωή του και εκποβισμό. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Κυρίε και κύριοι, τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλέ χώρε. Σε καταπλισμού προσφύγων, σε χώρε που τι έχει καταστρέψει ο πόλεμο, σε σοφρονιστικά ιδρύματα και αστυνομικά τμήματα, στου τάφους των δικών μου των φίλων, δημοσιογράφων, ακτιβιστριών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν ε, ε, δολοφονηθεί για να, τους, ε, για να τις φημώσουν η Νατάλια Σταμύροβα ε, και μία άλλη γνωστή μου δημοσιογράφη και ακτιβίστη ανθρωπίνων γυναικών που έχω συνάντησε στον πρώτο πόλεμο τη Τσετσενία στα ταξίδια μου, έκαναν κάτι που ονομάζω Δημοσιογραφία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα μείγμα τη αφήγηση με τη στήριξη των όσων αφηγούνται την ιστορία για να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά του και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το 2006 η Άννα Πολιτικόφσκα δολοφονήθηκε στη Μόσχα ε, στο ασανσέρ του, της πολυκατοικίας της τη μέρα των γενεθλίων του Πούτιν. Αυτοί που την δολοφόνησαν την Άννα ήξεραν ότι είχαν εγγυημένη ατιμορρησία. Δεν θα βρίσκονταν ποτέ. Αυτός που έδωσε την εντολή για την δολοφονία βέβαια ούτε καν. Αυτό συνέβη και με πολλούς άλλους δημοσιογράφους και ακτιβίστε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία πριν από την Άννα. Η Νατάλια Στεμίροβα, η οποία εργαζόταν ε, για την Μεμοριαλ Ρωσική ε, Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έκανε ανακριτική δημοσιογραφία για το τι συνέβαινε στην Τσετσενία. Απήχθη μπροστά στα σπίτι φίλη τη και δολοφονήθηκε στι 15 Ιουλίου 2009. Κανεί δεν έχει κατηγορηθεί για αυτό το φόνο, όπω και στην περίπτωση τη Άννα. Η Νατάλια έδειχνε τη βία μεταχείριση είχαν οι ε, άμαχε γυναίκε στην Τσετσενία από τι ρωσικέ δυνάμει και του ε, αξιωματικού τη Τσετσενία που χρηματοδοτούν οι Ρώσοι. Μέχρι τώρα οι αρχέ τη Ρωσία δεν έχουν καμία διάθεση να δουν ποιο έδωσε την εντολή για αυτέ τι δολοφονίε και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ένα χρόνο μετά το, τη δολοφονία τη Άννα, ε, ξεκίνησε ένα, την απονομή ενός ετήσιου βραβείου στο όνομά της, το βραβείο Ανά Πολιτικόφσκα. Ε, έχουν περάσει 7 χρόνια και σήμερα το βραβείο ε, φέτος θα το πάρει το βραβείο, μια ακτιβίστρια δημοσιογράφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω η Άννα ύψωσε το ανάστημά τη και μίλησε για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Νατάλια Στεμίροβα ήταν η πρώτη που κέρδισε το βραβείο Φυσικά το 2007 μέσα από αυτή τη δουλειά και με το βραβείο αυτά τα τελευταία 10 χρόνια μετά τη δολοφονία της Άννας Πολιτικόφσκα έχω συναντήσει μια ομάδα ε, εκπληκτικών γυναικών οι οποίες έχουν τιμηθεί με το βραβείο Άννα Πολιτικόφσκα και από το Αφγανιστάν ως το Ιράκ, από τον Ταρφούρ ως τη Συρία, οι γυναίκες που διακινδυνεύουν, ρισκάρουν τη ζωή τους για να πούν την αλήθεια, να σώσουν και να στηρίξουν τους αμάχους αυτές τις ενόπλες συγκρούσεις, πρέπει να τιμηθούν. Το 2011 νικήτρια ήταν η Ραζάν Ζάουτουμεκ από τη Συρία. Μια άλλη τολμηρή νεαρή γυναίκα η οποία τόλμησε να, να ψώσει τη φωνή της και να πει τις φρικαλαιότητες που ζει ο λαός της. Η πυγμή της να πει την αλήθεια, την ανάγκασε βέβαια να κρυφτεί στη συνέχεια και, την, ε, ε και επίσης και βασανίστηκαν τα μέλη της οικογένειάς, της. Οικογένειάς της. Ναι, ναι, ναι, θα κλείσω. Όμω συνέχισε την προσπάθειά τη από την κρυψώνα τη, από το κρυσφύγητό τη και για να αναγνωρίσουμε το κουράγιο του Δεκέμβριο του 2011, η Ραζάν έλαβε και το βραβείο Ζαχάροφ του, Ηνωμένου, του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, μετά η Ραζάν μαζί με δύο ακτιβίστε με τι οποίε συνεργαζόταν απήχθησαν από μέλη τη αντιπολίτευση και από ένοπλες Ισλαμιστικές ομάδες ε, και σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμη πού βρίσκονται. Η ιστορία απλώ επαναλαμβάνεται από την Τετσενία ως την Συρία και την Ρωσία περνώντας από τις ένοπλες συγκρούσεις των χωρών της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας τι βλέπουμε, οι δημοσιογράφοι, οι ε, πληροφοριοδότες, οι ακτιβίστριες ε, φυλακίζονται και δολοφόνονται όπως η Νατάλια και η Άννα γιατί δεν θέλουν να θυμωθεί η φωνή των γυναικών. Διαρκώ αναρωτιέμαι πώ μπορούμε να προστατεύσουμε αυτού που ακόμη τολμούν να μιλούν ε, κατάφατσα μπροστά στου κινδύνου. Θα πρέπει ε, να μην είμαστε αδιάφοροι, θα πρέπει να στηρίξουμε του δημοσιογράφου, συντάκτε, ε, ακτιβιστέ που δίνουν φωνή σε αυτούς που κανείς δεν θα άκουγε αλλιώ. Και πολύ σύντομα να πω ότι είναι πολλά αυτά που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Μην επικεντρώνεσαι μόνο στι γυναίκε ω θύματα. Να αναθεωρήσετε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και τι κατευθυντήριε γραμμέ για του υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να δώσετε ειδική προσοχή στι ανάγκε και την προστασία των γυναικών που είναι ε, ακτιβίστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίω αυτέ που εργάζονται σε χώρε ε, καταστάσει ενόπλων συγκρούσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ταχύ και αποτελεσματικό μηχανισμό για την προστασία του. Να θεσπιστεί ένα ειδικό καθεστώ θεωρήσεων για τι γυναίκε υπερασπίστε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να μπορούν να αποφέρουν σε έκτακτες συνθήκες τις απειλές και να σώζονται. Να ακούγεται τη φωνή τους και εδώ, η φωνή των γυναικών που είναι ακτιβίστες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει ένα μόνιμο συμβουλευτικό σώμα στη δική σας επιτροπή ή παρά τη για τις ε, γυναίκες υπερασπίστες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, συμπεριλαμβανομένων αυτών των χωρών σε ένοπλε συγκρούσει και από τις χώρες Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, για να μπορεί να ακουστεί η φωνή τους και να επηρεάσουν τις ε, πολιτικές προτάσεις για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θεωρήσετε τα μέσα χρηματοδότησης και τους μηχανισμούς, ώστε να υπάρχει στοχευμένη χρηματοδότηση για το έργο των γυναικών που είναι υπερασπίστες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την ειδική τους προστασία. Να αντιμετωπιστεί η, ατιμερο... η, η ατιμορρησία, η λογοδοσία είναι σημαντική για την προστασία των γυναικών και των θυμάτων βίας, βίας που έχει γίνει λόγω τη συνδικατική μεταχείριση λόγω φύλου, αλλά και στην περίπτωση των ε, συνομιλητών τη ειρήνη, των πληροφοριδοτών, των ακτιβιστριών, των δημοσιογράφων. Μην αφήνετε τη γυναική φωνή να φημώνεται. Σα ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σα. Σα ευχαριστούμε, κυρία Κατσάροβα. Σας ευχαριστούμε που μας μεταφέρατε την εμπειρία σας, τα μηνύματα που δώσατε, τις προκλήσεις που μας περιγράψατε, που είναι ακόμη τεράστιε. Και μας δώσατε μία η επισκόπηση της κατάστασης. Περάσαμε από τις γυναίκες στη θέση λήψη αποφάσεων, από την ανάγκη οικονομικής χειραφέτησης. Μιλήσατε για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη των σειράξεων και στο θέμα της ε, εξασφάλισης και διατήρησης ειρήνης. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία ε, Βερόνικα Ξεμπάλσκα, κοινωνιολόγο από την, Ευρωπαϊκή, από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών. Η κυρία Κρεμπάλσκα θα μας μιλήσει για τις πολιτικές που δεν συνάδουν με την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Γεια σας και ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή των Γυναικών για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα των κινητοποιήσεων ε, ε, για τις, κατά των πολιτικών που δεν συνάδουν με την ισότητα των φύλων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες επιτακτικές προκλήσεις ε, που εμφανίζονται και στην ανατολική εταιρική σχέση με την αυξανόμενη στρατοκρατία που μας ανέφερε η Μαριάννα, το μιλιταρισμό και η... τα κινήματα κατά της ΣΟΤΕΣ ε, δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις ε, και για τι χώρε Ανατολική Εταιρική Σχέση, αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών ακόμη και στο επίκεντρο, στην καρδιά τη Ευρώπη. Επίση, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή την πρόκληση δεν μπορούμε να την ε, αντιμετωπίσουμε με τις ε, συνήθεις ε, πολιτικές μας, με τις οποίες νιώθουμε άνετα. Για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις μας και να περάσουμε τις απλές πολιτικές, να ασχοληθούμε με την πολιτική με πει κεφαλαίο. Έχουμε πολλές συστάσεις πολιτικής που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η έκθεση αναφέρεται σε δύο βασικές προκλήσεις. Η πρώτη είναι η παραδοσιακή φαλοκρατούμενη, ανδροκρατούμενη κοινωνία. Εκεί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παραδοσιακές προκαταλήψεις, τα στερεότυπα ε, τη, για τη συμμετοχή των γυναικών, την οικονομική τους χειραφέτηση και την κοινωνική τους κατάσταση. Δεύτερη πρόκληση είναι το νομοθετικό σύστημα. Η, η ισότητα των φύλων δεν εξασφαλίζεται νομοθετικά στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Θα πρέπει να εφαρμοστούν και άλλα μέτρα. Σήμερα όμως εγώ δεν θα σας μιλήσω για τους συνήθει υπόπτου, δηλαδή την φαλοκρατούμενη, ενδροκρατούμενη κοινωνία και τα ε, φαλοκρατικά στερεότυπα και προκαταλήψεις ε, ή τα νομοθετικά μέτρα που είναι απαραίτητα. Θα επιστήσω την προσοχή σας σε μια, καινούργια πρόκληση που είναι τα πολιτικά, κοινωνικά και σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών που αρχίζουν και αυτά να φτάνουν στην ανατολική εταιρική σχέση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, διασυνοριακές ε, κινητοποίησεις ε, για να καταπολεμήσουμε τέτοιες πολιτικές που δεν συνάδουν την ισότητα των φύλων. Τα τελευταία τρία χρόνια ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Εγώ θα σας μιλήσω πρώτα εν συντομία για το τι γνωρίζουμε ήδη για τα κινήματα anti-gender. Μετά θα σας δώσω κάποια παραδείγματα των δραστηριοτήτων τους στις χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης και θα ολοκληρώσω με κάποια συμπεράσματα για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Τι είναι λοιπόν αυτά τα κινήματα anti-gender, γιατί ίσως δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με την έννοια αυτή. Πρόκειται για διασυνοριακά κοινωνικά κινήματα που κινητοποιούνται κατά των εχθρών της ιδεολογίας του φύλου, ε, της θεωρίας του φύλου και αυτό συμβαίνει και κυρίω ε, κυρίως ε, στις ανατολικές χώρε Ανατολική Εταιρική Σχέση. Ε, Στόχο του είναι τα δικαιώματα των γυναικών, ε, η συνεκτίμηση του φύλου, η ισότητα των φύλων, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι μελέτε για το φύλο ω ε, τμήμα του πανεπιστημιακού προγράμματο και διάφορε πρωτοβουλίε δικαίου σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Η έννοια του φύλου είναι συμβολική κόλλα, όπως είπε ένας στοχαστής, γιατί φαίνεται ότι δια, συγκεντρώνει διαφορετικούς συντηρητικούς παράγοντες υπό ένα κενό, κοινό όνομα, προκειμένου να ε, υπονομεύσει το ευρωπαϊκό σχέδιο, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα μέσα που βρίσκονται στην καρδιά των δημοκρατικών πολιτικών, δηλαδή κινητοποίηση στη βάση, δημοψηφίσματα και τις ε, ακτιβιστικές με κυβερνητικές οργανώσεις. Και παρόλο που τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, αυτή η κινητοποίηση κατά των πολιτικών ισότητας των φύλων, ε, τέτοιες κινητοποίησεις θα πρέπει να ε, κληθούν ω ε, τμήμα του διακρατικού διασυνοριακού φαινομένου και όχι ω τοπικά φαινόμενα. Υπάρχουν πολλέ διασυνδέσει μεταξύ διεθνών φορέων, καθώ και μεταφορά τεχνογνωσία, γνώσης και πρακτικών μεταξύ του. με αποτέλεσμα να καταλήγουμε σε μερικά κοινά χαρακτηριστικά αυτών των κινημάτων. Τώρα θα σας μιλήσω για αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι κοινή ανθρωπολογική βάση όλων των κινημάτων κατά των, της των φύλων. Ξεκινάνε από τα βασικά διδάγματα της Ρωμακοθαλικής Εκκλησίας. Ένα βασικό στοιχείο που στηρίζει τέτοιες ε, οργανώσεις είναι μια, ένας νέος ευαγγελισμός, ένα, το νέο Ευαγγέλιο των Χριστιανών ε, που ήδη είχαν ε, ασπαστεί τον χριστιανισμό. Επίσης, νέα διδάγματα για τις γυναίκες, για τη θέση τους στην κοινωνία, για, τη, για το σώμα των γυναικών και την ιδέα της συμπληρωματικότητας των φύλων. Γιατί οι γυναίκες και οι άνδρες είναι διαφορετικές, αλλά συμπληρώνονται τα δύο φύλλα. Δεύτερο χαρακτηριστικό αυτών των κινημάτων είναι ότι συμμετέχουν σε αυτά παρόμοιοι παράγοντες. Για παράδειγμα, βασικός παράγον είναι η Ορθόδοξη ή η Ρωμακοθολική Εκκλησία. Δεύτερος παράγον είναι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, European Dignity Watch ή το Ευρωπαϊκό Κογκρέσο Οικογενειών. Και μάλιστα πρόσφατα και στη Γεωργία έγιναν τέτοια πάνελ με ε, θέμα την, το, τον επικίνδυνο χαρακτήρα τέτοιες ιδεολογίες. Και κάποιες, κάποια πολιτικά κόμματα για να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους χρησιμοποιούν αυτό το θέμα της πολιτικής κατά της των φύλων. Επίσης έχουμε το, στη Γεωργία το ε, κίνημα των Ορθόδοξων οικογενειών και στην Ουκρανία κάτι αντίστοιχο. Έχουμε κινητο... τέτοιε κινητοποιήσει που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Χρησιμοποιούν κοινή φρασεολογία προκειμένου ε, να ε, μιλήσουν για την αξιοπρέπεια και, και το αίσθημα τη ασφάλεια, που είναι ένα θέμα προσφυλέ στον κόσμο. Έχουμε όμω ένα νέο απεικιοκρατικό πλαίσιο που χρησιμοποιούν αυτά τα κινήματα και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρουσιάζεται ως ο νέος επικιοκράτης και η ιδέα του φίλου ως απολυταρχικό ιδεολόγημα που καταστρέφει ε, τον τοπικό πληθυσμό εξυπηρετώντας τις εθνικές ελίτ. Και μέχρι στιγμή το κίνημα αυτό συγκεντρώθηκε στην, επικεντρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή θεωρεί ως εχθρό. Και οι πληροφορίε χώρε Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι ελάχιστε. Ναι, ξέρω, μιλάω πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, συνήθω μιλάω πολύ γρήγορα. Όπως είπα λοιπόν, η, μέχρι στιγμής ε, η έρευνα επικεντρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρουμε και πολλά για αυτές τις ε, διεθνείς ή διασυνοριακές κινητοποίησεις ε, στα, στις χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Παρόλο που ακτιβιστές από την Αρμενία, Ζαρβαϊζάν, Λευκορωσία, Μολδαβία και Ουκρανία έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου στη διεθνή κοινότητα για την ε, όλο και μεγαλύτερη αρνητικότητα και εχθρότητα απέναντι στο φεμινισμό, δεν υπάρχουν διεθνείς έρευνες για το θέμα αυτό. Οπότε ε, μπαίνουμε στην παγίδα να θεωρήσουμε ως τοπικά φαινόμενα τέτοιου είδους κινητοποίηση και όχι τμήματα ενός διακρατικού διεθνούς φαινομένου. Βέβαια μπορούμε να διασυνδέσουμε κάποια φαινόμενα στις χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με αντίστοιχες κινητοποίησεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν στις χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης βλέπουμε ότι συμμετέχουν παρόμοιοι φορείς όπως και σε άλλες χώρες. Η Εκκλησία, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κατά των αυλώσεων ή ε, ακροδεξιές οργανώσεις που έχουν διασυνδέσει και με τοπικά δίκτυα. Στη Γεωργία η Εκκλησία πρωτοστατεί σε τέτοιες ε, κινητοποίησεις κατά της ισότητας και βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη παρουσία εξτρεμιστικών ομάδων. Πρόσφατα είχαμε την επίθεση μιας την ε, ε, επίθεση κατά μιας καθετερίας στην Τυφλίδα, ε, ευρωπαϊκής και φεμινιστικής. Και το θέμα της, του αυξανόμενου μιλιταρισμού, της στρατιωτικοποίησης και στρατοκρατίας, και αυτό επιδίνωσε την κατάσταση. Για παράδειγμα, είχαμε απειλές κατά ε, ΛΟΑΔΜ σε μια εκδήλωση που έγινε σε ένα ξενοδοχείο. Χρειάζεται να κενωθούν με ειδική αποστολή και ειδικό λεωφορείο. Χρησιμοποιούν οι ομάδες αυτές τον εκφοβισμό και υπερβολική φρασιολογία και μάλιστα ε, μιλούν για σεξουαλικές ανομαλίες και παθολογίες κοινωνικές ε, προσπαθώντας να ξεσηκώσουν κατά των, ε, κόμμα κόμματος. Επίσης στην Ουκρανία είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο που θεωρούν ότι τέτοιου είδου ε, ισότητα των φύλων μπορεί να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα και να υποδουλώσει την Ουκρανία όπως είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση. Επίσης, ε, είπαν ότι η Ουκρανία προσυπογράφοντας το δίκαιο ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει θύμα της μετασοβιετικής μετακομμουνιστικής δικτατορίας. Έτσι έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κίνημα αυτό σύμβολο αυτής της, της πολιτικής. Και άλλες χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης από, ακολουθούν παρόμοιες δράσεις και παρόμοια ιδεολογήματα. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, κινητοποίηση στη Γεωργία, Αρμενία και Ουκρανία ξεκίνησαν με, την με, με το πρόσχημα της εφαρμογής κοινοτικών διατάξεων. Και στη Γεωργία μια εκδήλωση All Different All Equal ε, με διοργάνωση του, του Συμβουλίου της Ευρώπης προσέκρουσε στην αντίθεση της ε, εκκλησίας κατά μειονοτήτων και ε, φιλοευρωπαϊκών πολιτικών. Και στην Αρμενία ξεκίνησε μια τέτοια αντιτζέντερ εκστρατεία όταν υιοθετήθηκε η νομοθεσία για, τις, ε, για τα ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τους επόμενους μήνες ακροδεξιές ομάδες, ε, ε, συντηρητικοί και μη κυβερνητικέ οργανώσεις κατά της άβλωσης αποκάλεσαν τέτοιους ακτιβιστές ως εθνικούς προδότες και ανθρώπους που υπονομεύουν την οικογένεια. Ήταν πολλοί φορεί σε μέσα μαζική ενημέρωση και έγιναν πολλέ εξτρεμιστικέ οργανώσει, απειλώντα οργανώσεις ακτιβιστές ε, και ηθήνοντε για τη λήψη αποφάσεων. Η Ουκρανία είναι, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία περί ε, ισότητας, η πιο προηγμένη χώρα της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Και εκεί όμως έγιναν απειλές ε, με το πρόσχημα ότι απειλούνται οι ουκρανικές αξίες. Ξεκίνησε μάλιστα και μια εκστρατεία, το Stop Gender στην Ουκρανία. Ε, ξεκίνησε και μια πλατφόρμα στο ίντερνετ ε, με το ίδιο όνομα. Προωθήθηκαν βίντεο κλιπ στο ίντερνετ, μοιράστηκαν φυλάδια και ε, επιστολές προς τις ρωσικές και ε, ουκρανικές αρχές με στόχο τον εκφοβισμό των φορέων υπέρ της ισότητας. Τι ε, συμπεράσματα λοιπόν μπορούμε να συνάγουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα anti-gender κινήματα. Καταρχήν, αυτά τα κινήματα είναι μια νέα μορφή αντίσταση στην αλλαγή. Τέτοιου είδου ε, κινητοποίησει ε, χρησιμοποιούν νέα αφήγημα, νέε φρασιολογίε, νέα κινητοποίηση και περιλαμβάνουν και νέου φορεί και παράγοντε. Θα πρέπει να εκλειφθούν ω μια νέα πολιτική πρόκληση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παλιά μέσα. Άλλωστε, η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει τα δικά τη χαρακτηριστικά, τι ειδικέ τη ιδιαιτερότητε λόγω του ιστορικού και πολιτιστικού παρελθόντο. Και αυτό τα κινήματα αντιτζέντερ στι χώρε αυτέ κινητοποιούνται σε ένα πολύ χαλαρά οργανωμένο φεμινιστικό κίνημα και πολύ ισχυρέ φαλοκρατικέ και παραδοσιακέ αντιλήψει. Μάλιστα στην Αρμενία το 2010, 60% των ανδρών θεωρούν ότι οι γυναίκε δεν είναι κατάλληλε ηγέτηδε και πολλές γυναίκες, 60% των γυναικών λυπάται που δεν γεννήθηκαν άνδρες. Αυτές, οι προκαταλήψεις δημιουργούν μια παράδοξη κατάσταση που γυρίσει μπούμεραγκ στο φεμινισμό χωρίς να έχει διαπιστωθεί πραγματικά φεμινιστικό κίνημα πολλές εκδηλώσεις ε, κατά, το, του φύλου, κατά τις φύλου έχουν οργανωθεί στις χώρες αυτές, σε αντίθεση με φεμινιστικές που δεν οργανώνονται. Πρόκειται για διασυνοριακά φαινόμενα και κινητοποιήσεις που έχουν και τοπικές εκφάσεις, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλα τα επίπεδα, και τοπικό και διασυνοριακό. Και όπως είπε και ο Ανδρέα Πέτσαλ, μια προοδευτική ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να ξεπεράσει το γραφείο, τη γραφειοκρατική της εστίαση στην εφαρμογή των πολιτικών και της ρύθμισης. Θα πρέπει να επιστρέψει στα αίτια, στη βάση και θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότερες προσπάθειες για να στηριχθούν τοπικές ομάδες, οργανώσεις και πρωτοβουλίες που θα δώσουν την εναλλακτική λύση σε αυτές τις νεοσυντηρητικές ε, κινητοποίησεις τέτοιε ακτιβιστικέ ομάδε και ομάδε ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρήζουν όχι μόνο οικονομική αλλά και πνευματική υποστήριξη για να αντιληφθούν ότι προσπαθούν να αντιμετωπίζουν ένα διασυνοριακό φαινόμενο και όχι ένα τοπικό, φαλοκρατικό ή ανδροκρατούμενο μπούμεραγκ. Θα πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε πολλέ πρωτοβουλίε και σεμινάρια, γιατί τοπικοί ακτιβιστέ ε, γνωρίζουν ε, του φόβου και τον προβληματισμό του τοπικού πληθυσμού και μπορούν καλύτερα να αντιδράσουν και να βοηθήσουν του ηθήνοντε τη πολιτική να τα μεταφέρουν σε πραγματικέ πολιτικέ. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τη βάση και τι τοπικέ οργανώσει, Αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί όλο και περισσότεροι, όχι μόνο στι χώρε ανατολική Εταιρική σχέση, αλλά και στην Ευρώπη, γίνονται όλο και πιο σκεπτικιστέ κατά τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αρχίζουν και ε, αμφιταλαντεύονται για το κατά πόσο η πρόοδο αγγίζει όλου και, μόνο, και όχι μόνο ορισμένου. Γι' αυτό θα πρέπει να αναζωογονήσουμε τον ίδιο τον τρόπο σκέψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα. Και δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τα κινήματα αντιτζέντερ ως απλή αντίσταση στο φεμινισμό. Θα πρέπει να τα δούμε με το πραγματικό τους πρόσωπο. Είναι μια νεοσυντηρητική απάντηση σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα διασυνοριακής κρίσης παγκοσμιοποιημένης νεοφιλελεύθερης δημοκρατίας. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο τα κινήματα αντιτζέντερ προέρχονται από τους φόβους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, τον αφιλελεύθερο οικονομικό καθεστώς και τις αποτυχημένες ε, υποσχέσεις ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μετά προβάλλονται στο, στο θέμα στο ρόλο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι σημαντικό λοιπόν να κινητοποιηθούμε για την ισότητα των φύλων, προσπαθώντα να χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού και τα αίτια στη βάση. Θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα των ε, εκκλησιαστικών και ε, άλλων οργανώσεων κατά των αυλώσεων. Θα πρέπει να δώσουμε μια εναλλακτική λύση που θα ανακτά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι σίγουρη ότι η συνεισφορά σας ε, θα θέσει εκ νέου ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σημαντική οπτική γωνία που μας ε, δώσατε. Ε, έχω το δικαίωμα αργότερα να κάνω και ερωτήσει, πιστεύω. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Vincent Φόρεστ, ο οποίο είναι διευθυντής ε, παρεμβάσεων ε, υπέρ των δικαιωμάτων στην Ευρωμεσογειακή περιοχή και θα ασχοληθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, ε, τον ρόλο των γυναικών και τον τρόπο που η πολιτική αυτή συνεχίζει να προωθεί την ισότητα των γυναικών στις χώρες ε, της νότιας ε, γειτονίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Είμαι ο Vincent ε, Forrest από το Euromed Rights. Θα πω ότι καταρχάς χαίρομαι που θα συνεισφέρω στην ισότητα των φίλων σε αυτό εδώ το πάνελ. Θα χρειαζόμουν πολλές ώρες να μιλήσω αν μίλαγα αργά, γι' αυτό θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ. Να πω ότι το γύρο Med Rights είναι ένα δίκτυο με 70 οργανώσεις που έχουν τη βάση τους και στην Ευρώπη ε, και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι 50-50 λοιπόν, γιατί ε, έχει την ευρωμεσογειακή οπτική γωνία και συμπεριλαμβάνει και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Εγώ παρακολουθώ αυτή την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια και ειδικότερα την αναθεώρηση πέρυσι και την ανακοίνωση τη σχετική τον περασμένο Νοέμβριο. Και συγκεκριμένα έχουμε μια ομάδα εργασία με μεικτή σύνθεση. Η μισή είναι από την Ευρωπαϊκή η Ένωση, άλλη μισή από τις χώρες της νότιας γειτονίας. Όμως επικεντρωνόμαστε κυρίως στην κατάσταση στις νότιες χώρες, συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε στη βία κατά των γυναικών. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πως από, ε, κυρίως από τις εξηγέρσεις της αραβικές χώρες αλλά και πριν από αυτό είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις, νομοθετικές αλλαγές, προοδευτικά συντάγματα στο Μαράκο το 2011, στην Τινησία και την Αίγυπτο πριν από δύο χρόνια Ακόμα και πριν είχαμε την αναθεώρηση του οικογενειακού κώδικα στο Μαρόκα, έναν ε, ε, νόμο στην Αίγυπτο το 2008 για τον ακροτηριασμό των ε, γεννητικών οργάνων, ο οποίος απαγορεύτηκε. Το, στο Λίβανο επίσης το 2014 αντίστοιχε νομοθεσίες, όπως και στην Αλγερία. Και υπήρξαν και πιο συνολικοί νόμοι που πέρασαν φέτος στο Μαρόκο για την βία κατά των γυναικών, αλλά και στην Τινησία. Βέβαια υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτή την ομάδα εργασίας ε, για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, όμως στην ουσία έπρεπε να μιλάμε για ανισότητα των φύλων στην περιφέρεια αυτή, διότι οι περισσότερες χώρες έχουν κυρώσει την αντίστοιχη σύμβαση, αλλά έχουν επιφυλάξεις για πολλά άρθρα, εκτός από την Τινησία που ε, κατάφερε να τις επιφυλάξεις, αλλά υπήρξαν και άλλες χώρες ε, που ε, πριν από δύο χρόνια υπέγραψαν χωρίς επιφυλάξεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θετική στροφή σε νομοθετικό επίπεδο, όμως πολλές από τις νομοθεσίες έχουν πολύ περιορισμένο πεδίο. Για να απαντήσω και στο ερώτημά σας σχετικά με το χάσμα ανάμεσα στην, κοινότητα, στην κοινωνία συγγνώμη, των διαφόρων χωρών και τη νομοθετική παρέμβαση να πω ότι οι νόμοι συνήθως αντικατοπτρίζουν τις συντηρητικές ε, αξίες οικογενειακές και όχι τις προοδευτικές ε, τάσεις. Να πω ότι το 2008 είπαμε ότι στην Αίγυπτο ε, εγκρίθηκε ένας νόμος κατά του ακροτηρισμού των γεννητικών οργάνων. Παρόλα αυτά, μια κοπέλα 17 πέθανε το Μάιο ε, μετά από επιπλοκές ε, λόγω αυτής ε, της επέμβασης ακροτηριασμού. Φαίνεται λοιπόν ότι η νομοθεσία τελικά δεν έχει φέρει το τέλος σε αυτή την πρακτική. Ήταν απλώς μία αρχή και το πιο σημαντικό είναι να δούμε την εφαρμογή και την πράξη. Υπάρχει και μια μεγάλη άλλη πρόκληση, αυτό που είπε η Μαρία πριν. Οι γυναίκες ε, η Μαριάννα μάλλον, ε, οι γυναίκες ε, δεν στιγματίζονται επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επειδή είναι γυναίκες. Έχουν λοιπόν συνεχώς απειλές να αντιμετωπίσουν που έχουν να κάνουν με το φίλο τους και με το γεγονός ότι προσπαθεί κανείς να μειώσει την αξία του έργου τους. Γενικά αυτό γίνεται σε όλες αυτές τις χώρες. Οι συνάδελφοί μου που είναι ε, που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα μιλάνε ε, για το πώς ε, έχει δημιουργηθεί ένα μπούμεραγκ διότι Υπάρχει ένα αυτή η θετική τάση με την νομοθεσία, όμως οι γυναίκες τελικά στοχοποιούνται περισσότερο επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η νομοθεσία από διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Ε, κοιτώντας τώρα τα ε, διεθνή ε, μέσα και τα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέσο που να ασχολείται με την νότια πολιτική γειτονίας. Ε, ε, θα δούμε λοιπόν τα γενικότερα ε, μέσα. Έχουμε το σχέδιο δράσης για το φύλλο. Θα μιλήσει και η συνάδελφος μετά για το δεύτερο τέτοιο σχέδιο δράσης. Έχει γίνει μια συστηματική λοιπόν ανάλυση για όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το όλο και περισσότερο στη μετάφραση των λόγων σε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Θα δούμε τι θα γίνει, σημαίνει αυτό ε, επιτόπου. Ε, ξεκινώντας όμως με τις συστάσεις να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ξεκάθαρο μηχανισμό παρακολούθησης ε, για να δούμε πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη ας πούμε το σχέδιο δράσης για το φύλλο γιατί ξέρουμε ότι στην πρώτη του εκδοχή υπήρχαν κάποια προβλήματα κυρίως ε, στο θέμα της ε, ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλλου. Γι' αυτό λοιπόν, όπως μόλις είπα, οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που απονομιμοποιούνται είναι κάτι στο οποίο ε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ε, να προστατεύουμε δηλαδή τα άτομα, ε, να έχουμε ευρωπαϊκές οδηγίες για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη βία κατά των γυναικών. Στην αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία υπάρχει μια αναφορά στο σχέδιο δράσης για το φύλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αντιμετωπίζονται τα, δικαιώματα των γυναικών Τώρα με το Λίβανο, την Ιορδανία και την ε, Αίγυπτο και σύντομα με την Αλγερία θα υπάρξει μια προσέγγιση και έχω ακούσει ότι εκεί τα δικαιώματα των γυναικών θα αποτελέσουν προτεραιότητα της εταιρική σχέσης και ένα θέμα που θα διατρέχει όλους τους τομείς. Το σημαντικό γενικά είναι το φύλλο να αποτελεί ε, βασικό σημείο των πολιτικών, των προτεραιοτήτων αλλά και της εφαρμογής τους ε, ε, και, των εκθέσεων επί της εφαρμογής τους. Επίσης είναι σημαντικό και κρίσιμο ε, όποια βήματα γίνονται υπέρ των γυναικών να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με το Μαρόκο ας πούμε και την Τινησία. Είδαμε πρόσφατα νομοθεσίες που πέρασαν αλλά το περιεχόμενό τους ε, δεν ήταν ικανοποιητικό. Ε, υπάρχουν δηλαδή ε, άρθρα τα οποία αποδυναμώθηκαν πριν περάσουν. Υπάρχουν πολλές λοιπόν προκλήσεις. Θα τελειώσω όμως με μία αναφορά στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών. Γιατί, Γιατί είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο, εργαλείο και αρκετά ολοκληρωμένη κάλυψή του. Βέβαια είναι ανοιχτό προσκύρωση όχι μόνο από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και από άλλα μέλη ε, μεταξύ αυτών και των ε, νότιων μεσογειακών χωρών. Υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την κύρωση. Να σας πω ότι το φθινόπωρο θα ξεκινήσει και μια δημόσια εκστρατεία για τη σύμβαση για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών, γιατί δεν υπάρχει γνώση, δεν, υπάρχει, ε, δεν είναι ορατή η σύμβαση και θέλουμε να επηρεάσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις για να εφαρμόσουν, όχι μόνο να προσυπογράψουν και να κυρώσουν, να εφαρμόσουν και τις διατάξεις. Έχουμε τα τέσσερα π. προς, ε, η προστασία, πρόληψη ε, και οι ολοκληρωμένες πολιτικές. Υπάρχουν έξι χώρες, η Γαλλία, η Κύπρος, η Τουρκία, στο βορρά, Μαρόκο, την Ισία, η Ορδανία στο νότο. Ε, οι τρεις στο νότο δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη σύμβαση. Η Κύπρος έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει. Η Γαλλία και η Τουρκία μόλις ε, κύρωσαν και τώρα έθεσαν σε ισχύ. Γιατί η Γαλλία και η Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλά ε, μειονεκτήματα. Ας πούμε στη Γαλλία υπάρχει ατιμορρησία. Λιγότερες είναι οι καταδικαστές αποφάσεις σε σχέση με τις ε, προσφυγές. Ε, έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα εξ αρχής, ε, να έχουμε αυτή τη διάσταση την ευρωμεσογειακή και να μην μιλάμε μόνο σε συναδέλφους και κυβερνήσεις ε, στο Νότο, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, να πω ότι έχω φέρει ε, αντίγραφα του δελτίου σχετικά με τις διάφορες χώρες. Υπάρχουν ε, αυτά τα αντίγραφα διαθέσιμα στην γραμματεία για την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, το Μαρόκο και την Τινησία που περιγράφουν την κατάσταση, την νομοθεσία και δίνουν δεδομένα και αριθμούς για αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ και σταματώ εδώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Φόρες, ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με τις ε, χώρες της νότιας πολιτικής γειτονίας και τώρα φτάνουμε στην τελευταία ομιλήτρια η οποία ήδη ε, σε προηγούμενες παρεμβάσεις υπέστησε ερωτήσεις γιατί είναι η κάθε φορά που αναφέρεται η Κομισιόν, σε εσά πέφτουν τα βλέμματα. Η κυρία Έμα Σαντάλ, διεθνής αξιωματούχο για την ε, βοήθεια και τη συνεργασία από την Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡΑ, της γειτονίας και της διεύρυνση δηλαδή, και ε, θα μας μιλήσει για τις δυνατότητες που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και για τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, αυτό το θέμα, το χρηματοδοτικό, πρέπει να το συζητήσουμε για την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών. Επίση. είστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του νέου σχεδίου δράση για το φύλλο, που αναφέρθηκε ήδη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η παρακολούθηση. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την παρέμβασή σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση η Γενική Διεύθυνση NEAR που καλύπτει τις, ε, ε, και την Ανατολική και την Νότια γειτονία αλλά και τις χώρες της διεύρυνσης ε, έχει μεγάλη δέσμευση, θέλει να προχωρήσει στο θέμα της ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης των γυναικών ε, τα επόμενα χρόνια ε, στις γειτονικέ χώρες. Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας που αναφέρθηκε δίνει έμφαση στην ισότητα των φύλων αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες, τις κοινωνικές και τις υπηρεσίες δικαιοσύνης. Επίσης, η πάταξη των ανισοτήτων είναι κομμάτι της προσπάθειας να προλάβουμε την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση. Το Ευρωπαϊκό ε, Σχέδιο Δράσης για το Φύλλο 2016-2020 παρέχει ένα καλό πλαίσιο με το οποίο θα διασφαλίσουμε ότι τα καλά λόγια που λέγονται τελικά θα γίνουν και πράξη. Όπως αναφέρθηκε, το προηγούμενο σχέδιο δράσης για το φύλλο δεν ήταν ε, επαρκές. Δεν έφτανε μέχρι το τέλος και αυτό αναγνωρίστηκε όταν ξεκίνησε η εργασία μας και ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε στον GAP2, όπως το λέμε πλέον. Ε, μιλήσαμε για τη διαχείριση των πόρων, για την παρακολούθηση της εφαρμογής, το follow-up δηλαδή. Πήραμε κάποια μαθήματα και η διαδικασία αξιολόγησης ε, από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη-μέλη οδήγησε σε μια συζήτηση που μας έφερε στο GAP 2. Παρόλο που η κατάσταση των γυναικών διαφέρει στις διάφορες χώρες, υπάρχουν κοινά προβλήματα, υψηλά επίπεδα βίας κατά των γυναικών, σημαντική και η διαφορά ε, στι αμοιβέ των γυναικών σε σχέση με του άντρε και λιγότερη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ ε, που ε, υπάρχει μόνο 1,5 χρόνο πριν ήταν η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, θα τη λέω ΝΙΕΡ, έχει δώσει 103 εκατομμύρια ευρώ σε 111 προγράμματα που προωθούν την ισότητα των φύλων και την κατάσταση των γυναικών σε όλη την περιφέρεια, κυρίως στην νότια γειτονία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ ε, σε προγράμματα για τις γυναίκες και την επιχειρηματικότητα, διότι θέλουμε να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα των γυναικών και τη συμμετοχή τους στο επιχειρήν, δίνοντας πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στα υπηρεσίε ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Επίσης, έχουμε σχέδια για 5 ε, προγράμματα για τις γυναίκες των Ηνωμένων 13,8 ε, εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με την οικονομική και κοινωνική δυνάμωση των γυναικών στο Νότο και ε, τεχνική βοήθεια για την βία κατά των γυναικών. Επίσης αναφέρθηκε η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, π.χ. η Γεωργία που έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει. Επίσης ε, θα δοθεί υποστήριξη και στις τρεις θεματικές ε, ενότητες του Ευρωπαϊκού ε, Σχεδίου Δράσης, οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών, ψυχική και σωματική αγκαιρεότητα, η φωνή η χειρή φωνή για τις γυναίκες και συμμετοχή ε, των γυναικών. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Στην χρηματοδοτική υποστήριξη ε, που δίνουμε πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι προωθούμε την ισότητα των φύλων, ανδρών και γυναικών. Θέλουμε να αυξήσουμε την ε, συμμετοχή των γυναικών. Ε, όλες οι αντιπροσωπείες και οι μονάδες εδώ ε, εργάζονται επί της εφαρμογής της ΓΑΠ. Υπάρχει ένα σημείο μακαθοδήγησης που έχει εγκριθεί από το Γενικό Διευθυντή και μας συνδέει και πάλι με τις αποτυχίες της του GAP 1 που στην ουσία πλέον ε, μας οδηγεί σε καλύτερη υποστήριξη σε επίπεδο διαχείρισης. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, ένας τέταρτος τομέας ε, που κάποιος θα το έλεγε ε, ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αλλά στην ουσία είναι αλλαγή κουλτούρας. Επίσης, ε, το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα συνεχίσει να δίνει υποστήριξη για τις τρεις θεματικές ενότητες. Όλες οι αντιπροσωπείες κάνουν ανάλυση των φύλων. Αν ήδη δεν έχει γίνει λοιπόν, ε, θα έχουμε προγράμματα που θα είναι πιο καλά ενημερωμένα και θα περιλαμβάνουν και στατιστικές. Ήταν και ένα από τα ερωτήματα αυτό. Επίσης, Έχουμε ένα σύστημα τεχνική υποστηριξή για χώρε που καλύπτονται ε, από τα ΕΠΑ ή το ΕΝΗ. Το ΕΠΑ είναι προταξιακό, προταξιακό εργαλείο. Έτσι, είναι ένα σημαντικό σύστημα που βοηθά στην, στην ε, μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και προωθεί τη συνεργασία σε θεμελιώδεις ε, αρχέ και πολιτικέ. Σκοπός είναι να δώσει σε υποψήφιους και δυνητικούς υποψήφιους ε, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνογνωσία με οργάνωση εργαστηρίων, αποστολή εμπειρογνωμόνων ή ε, επισκέψεις μελετών ε, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη για την μεταρρυθμίση της, διοικητικής, της δημόσιας διοίκησης αυτών των χωρών. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε υποβολή αιτήσεων τα με θέμα την ισότητα των φύλων, ε, να προωθήσουμε μηχανισμούς ισότητας ε, φύλων και στήριξη του ΤΑΓΕΞ και να προσφέρουμε feedback και ιδέες σε δραστηριότητες για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων μέσω του ΤΑΓΕΞ και της ε, συνδρομής που προσφέρουμε μέσω του ΤΑΓΕΞ. Έχουμε και κάποια παραδείγματα σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΝΗ γυναίκες στις επιχειρήσεις, ε, ε, gender budgeting, ε, δημοσιονομική υποστήριξη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτη φορά που χρησιμοποιείται δημοσιονομικός μηχανισμός γι' αυτό. Και είναι ένα θέμα συναφές και με την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολος. Για τον Νότο είχαμε πολλά προγράμματα όπως οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών, βελτίωση της, της, του βιωτικού τους επίπεδου σε μειονεκτικές περιοχές στο Λίβανο, συμπερίληψη των γυναικών σε, στην ειρηνική μετάβαση, στη μετάβαση στην ειρήνη στη Συρία. Επίσης άλλα προγράμματα που ενισχύουν την ε, θέση των γυναικών σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο και μάλιστα η συνεκτήμηση διάστησης του φύλου απαιτείται σε όλα τα προγράμματά μας σε συνδυασμό με το πρόγραμμά μας για την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δείκτες ε, για το φύλλο. Είναι ο δείκτης OSA, DAC. Παρακολουθούμε συστηματικά τα προγράμματα και τα σχέδια και αν ο δείκτης είναι μηδενικός θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί δεν περιλαμβάνεται η διάσταση του φύλλου. Και ελάχιστα είναι αυτά τα προγράμματα που έχουν τέτοιο μηδενικό δείκτη. Και η κλίμακα περιλαμβάνει βαθμολογία 1 και 2 και χρησιμοποιούνται και ομαδοποιημένα στοιχεία, checklists, ε, ε, ποιοτικές αξιολογήσεις και επίσης στις επιτροπές με τα κράτη-μέλη το θέμα της ισότητας των φύλων ε, αναφέρεται τακτικά. Και η Γενική Διεύθυνση ε, αναφέρεται τα θέματα στους διαλόγους πολιτικής με κυβερνήσεις και εκπροσώπους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, γιατί η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών ε, είναι αναπόσπαστο στοιχείο του μηχανισμού και του ΙΕΝΑ και της πολιτικής γειτονίας. Χρηματοδοτούμε και μελέτες. Έχουμε χρηματοδοτήσει μελέτες, για παράδειγμα, για την συμπερίληψη των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να έχουμε καλύτερα εμπεριστατωμένα προγράμματα. Επίση, στηρίξαμε την ομάδα υψηλού επίπεδου που έγινε στη Τυφλίδα, στη Γεωργία, πέρυσι. Παρουσία τη ε, υπάρξη εκπροσώπου αντιπροέδρου Μογκερίνη, που ήταν και η κεντρική ομιλήτρια. Και έχουμε και εταιρική σχέση με, την, με, την, των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών και το θέμα των ε, βέλτιστων πρακτικών μα ενδιαφέρει. Προσπαθούμε να έχουμε ανταλλαγέ με τα κράτη-μέλη, άλλε γενικέ διευθύνσει, οργανώσει κοινωνία των πολιτών, οργανώσει ε, των Ηνωμένων Εθνών, τη Παγκόσμια Τράπεζα, για προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτούνται από το ENI, ε, από το σύστημα αυτό ή από άλλε γενικέ διευθύνσει. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί για να μάθουμε όλο και περισσότερα, να αντλήσουμε διδάγματα και να συγκεντρώσουμε εμπειρίες για καλά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές. Αυτά, αυτά προς το παρόν, μια και ο χρόνος πίεζε και περιμένω τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή σας την ε, εισήγηση. Ευχαριστώ ε, λοιπόν ε, για τις παρουσιάσεις σας και να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις. Κύριε Μπαστιά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πλούσια ενημέρωση που μας κάνατε. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί μιλάω ισπανικά. Ευχαριστώ θερμά για την πληθώρα πληροφοριών που μας δώσατε, για την παρουσία σας εδώ και κυρίως για την ευκαιρία που μας δίνετε να συντάξουμε, να εκπονήσουμε μια τέτοια έκθεση που πάνω απ' όλα θα πρέπει να είναι επικριτική και να αναγνωρίσουμε την κατάσταση των γυναικών στις χώρες και της Ανατολικής και της Νότιας εταιρικής σχέσης. Πρόκειται για χώρες με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς, είτε εταιρική σχέση, είτε σχέση στα πλαίσια της πολιτικής γειτονία. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που μας προβλημάτισαν και πολύ ανησυχητικά Μιλήσαμε για τον Νότο, Μαρόκο, την Ισία. Έχουμε μια προνομιακή εταιρική σχέση με το Μαρόκο, που μάλιστα χαρακτηρίστηκε παράνομη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν αποφασίσει ε, αρχικά να μην ε, εφαρμόσουν, να μην τηρήσουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να ε, την εφεσιβάλλουν. Και μάλιστα δρομολογείται και αντίστοιχη συμφωνία με την Τινησία. Πρόκειται για δύο χώρες στις οποίες η κατάσταση των γυναικών είναι καταστροφική. Αναφέρθηκε ο οικογενειακός κώδικας. Με τέτοιους οικογενειακούς κώδικες τι κάνουν οι χώρες του Μαγκρέμπ. Ουσιαστικά παλινδρομούν σε σχέση με το γενικό επίπεδο της νομοθεσίας και έτσι επιτρέπουν τις διακριτικές μεταχειρήσεις και τις διακρίσεις βάρος των γυναικών. Εγώ ως δημοσιογράφος είχα ε, μιλήσει με γυναίκες από το Μαρόκο ε, για τις οποίες ε, είχε, δοθεί, ε, είχε το καθεστώς του άσυλο γιατί ήταν θύματα βίας, βίας λόγω φύλου. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε τις συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες αυτές, στις οποίες καταπατούνται τα γυναικεία δικαιώματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες ως μοχλό για να προωθήσουμε κάποιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες συμφωνίες, γιατί αυτό είναι το μόνο κατασταλτικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, ο μόνος μηχανισμός για να πιάσουμε τις χώρες αυτές να εξυγχρονιστούν σε θέματα ισότητας φύλου. Άλλο ανισχυτικό πράγμα είναι κάτι που ακούσαμε από τη δεύτερη ομιλητρία που μας μίλησε για κάποια ε, διασυνοριακά κινήματα και κινητοποιήσεις ε, που προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτή την ιδεολογία του φίλου, τη ισότητα του φίλου και μιλούν για δικτατορία της ισότητας του φίλου και μάλιστα ταυτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τη θεωρούν ως ε, προτέτειο και φυσικό αυτούργο αυτή τη δικτατορίας ε, της ισότητας ε, του φίλου Και θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα του υποδουλώσει με αυτή την ιδεολογία. Αυτά θα ήθελα να ρωτήσω είναι πολύ ενισχυτικό. Μάλιστα και από τη Βαλέση, από τη γενέτειρά μου, ο επίσκοπος είχε αναφέρει κάτι τέτοιο πρόσφατα. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους κινήματα διασυνοριακά που είναι ολοκληρωτικά, πολυτερχικά, που ουσιαστικά θέλουν να διατηρήσουν την φαλοκρατική κοινωνία και να κρατήσουν υποβαθμισμένο το ρόλο της γυναίκας. Πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους κινήματα, πέραν τη συζήτηση που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτά. Θα καταθέσουμε τροπολογία στην έκθεση προκειμένου να ενισχύσουμε την πίεση που θα πρέπει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις γειτονικές χώρες μέσω των προνομιακών αυτών σχέσεων και μέσω της διεθνούς μας ίσως εμπορικής πολιτικής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να εξάρουμε τη σημασία που έχει αυτή η έκθεση και να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της συγκεκριτρίας να θεωρηθεί Πρώτη τάξη αυτή η έκθεση και να ληφθεί υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για τις χώρες γειτονία, αλλά και εντός της Ευρώπης, γιατί υπάρχουν ανταλλαγές πληροφοριών, υπάρχουν ανταλλαγές δυνάμεων, δεν είναι τελείως ξεχωριστά αυτά τα θέματα και στο μέτρο που δεν βελτιώνεται η κατάσταση ε, εκτός Ευρώπης δεν πρόκειται να βελτιωθεί και εντός θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το θέμα τη ισότητα όχι μόνο στι γειτονικέ χώρε, χώρε εταιρική σχέση, αλλά και στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σημαντικό αυτό που είπατε ότι η παρουσία των γυναικών είναι πολύ ασθενή στα ε, στις διαπραγματευτικές ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε και εμείς τη, τη δύναμη και την παρουσία και την εξουσία στις γυναίκες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν ε, τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας. Πολύ ενδιαφέρον θέμα να αφισβήτητα και δυστυχώς θα χρειαστεί να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο θέμα αυτό. Εγώ θα τονίσω μία πτυχή ε, της ε, τις συζήτησης αυτής ε, για τα δικαιώματα των γυναικών και κυρίως ε, στην πολιτική γειτονία και στις χώρες της εταιρικής σχέσης. Στο σημείο 8 αναφέρεται ότι καταδικάζει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες ε, υπόκεινται οι γυναίκες Σαχαραουή στα κατεχόμενα από το Μαρόκο εδάφη, κυρίως ε, στις διακρίσεις ε, σεξουαλική βία και μηχανισμού που χρησιμοποιούν οι κατεχόμενες δυνάμεις του Μαρόκου για να εμποδίσουν ε, τον νόμιμο και εύλογο γόνατο των Σαχαροϊτών για αυτοδιάθεση και άσκηση των δικαιωμάτων. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο εγκρίθηκε στην Ολομέλεια της Ένωσης για τη Μεσόγειο, ψήφισμα που μιλά για τη σημασία των γυναικείων οργανώσεων στην προσπάθεια καταπολέμησης ε, των παραβιάσεων αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γυναικείων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν, λέμε στην ε, Ένωση ε, για τη Μεσόγειο, να περιλάβουμε όλες τις μορφές βίας, ακόμη και αυτές που πορεύουν από, την ξένη, από τις ξένες δυνάμεις κατοχής στην περιοχή. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχουν ειδικά προγράμματα στήριξης των γυναικών της Παλαιστίνης ε, στη, στα παλαιστινιακά κατεχόμενα ή στήριξη των γυναικών ε, Σαχαραουή κατά της ε, κατοχής του Μαρόκου. Και όπως είπε και ο Τζόρτι, έχουμε πολύ σημαντικές εμπορικές συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιες χώρες με το Ισραήλ, με το Μαρόκο, θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό πίεσης για να πετύχουμε βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις τελευταίες δηλώσεις του Ερντογκάν για τις γυναίκες. Μάλιστα τη στιγμή που επιδεψιλεύουμε τεράστια κονδύλια στον Ερντογκάν για μια υπονείδηστη κατά τη γνώμη μου συμφωνία για τους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά να έχουμε ένα πολιτικό ορθό αφήγημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απ' την άλλη να ασκούμε πολιτικές που είναι τελείως αντιφατικές με αυτό το αφήγημά μας. Θα πρέπει να δείξουμε πυγμή, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα υποφεληθώ για να θέσω και εγώ τις ερωτήσεις μου. Μία ερώτηση και για τους τρεις σας για τους τέσσερις μάτων, εάν μία πρακτική έπρεπε να επιλέξετε στον τομέα ειδικευσής σας, ποια θα ήταν αυτή, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε για να την υποστηρίξουμε, να την προωθήσουμε. Είναι ερώτηση και για τους τέσσερις αγορητές. Επίσης μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για την κυρία Γκριμπάσκα. Πραγματικά εξεπλάγει με το πόσο διεξοδικά αναλύσατε αυτού του είδους τις κινήσεις, μου μένει μία ερώτηση. Για να πετύχουν αυτά σε επίπεδο της κοινωνίας, τι πρέπει να γίνει. γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν ενώ προκαλούν αντεπιχειρήματα δεν είναι αυτά όσο ισχυρά και τελικά δεν καταφέρνουν να πετύχουν αυτό που θέλουμε για τις γυναίκες. Και επίσης μία ερώτηση για τον κύριο Φορέ. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει η κοινοβουλευτική διπλωματία. Οι γυναίκες εκτός από τις ε, θέσεις εξουσίας, εκτός από τις θέσεις στη δικασία λήψη αποφάσεων, ε, μπορεί να έχουν θέσει και στο Κοινοβούλιο, <clears throat> στην Τινησία, στο Μαρόκο, στην Ανατολική Γειτονία. Πώς μπορεί αυτή η κοινοβουλευτική διπλωματία να συμβάλλει για να προσπιστούμε καλύτερα τα δικαιώματα των γυναικών. Και έχω και μία ερώτηση για τη μετανάστευση. Κατεξοχήν θέμα επικαιρότητα. Έχουμε στοιχεία Κυρίω εδώ ε, απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ποσοστά μετανάστευση κάποιων χωρών, διότι οι λίγες πληροφορίες που διαθέτουμε ε, υποδεικνύουν ότι είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά μετανάστευση. Ποιοι λόγοι μπορούν να, τις εξηγήσουν, να τα εξηγήσουν αυτά, θα μπορούσε να υπάρξει αντιστροφή των γενεσουργών αιτίων. Υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ αυτών των χωρών που οδηγεί προ την ε, μετανάστευση προ το εξωτερικό και μετά για την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση. Συνεχίζει να είναι ένα από τα βασικά σημεία που σα απασχολούν και όταν μιλάω για την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση δεν εννοώ τα δευτεροβάθμια ή την πρωτοβάθμια, εννοώ την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή πώ πάνε οι γυναίκε στα πανεπιστήμια, ε, ισότητα των φίλων έχει να κάνει και με αυτό το στοιχείο κλειδί λοιπόν, την εκπαίδευση. Ήθελα την άποψή σα και για το θέμα αυτό. Και τώρα να δώσω πάλι το λόγο στους προκεκλημένους μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Κυρία Κατσάροβα, να δώσω πρώτα το λόγο σε εσάς. για την ερώτησή σας για τα θετικά παραδείγματα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι στο χώρο της ειρήνης, των συνομιλιών ειρήνης και την πρόσβαση των γυναικών στα τραπέζια των δημοτεύσεων, πρέπει να αναγνωρίσουμε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία των πολιτών και τον ρόλο της και τις ομάδες των γυναικών. Έχει πραγματικά υπάρξει ευρωστότατη αυτή η, κοινο, κοινωνία των πολιτών, θαλερή στις περισσότερες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Έχουν υποστεί διώξεις, έχουν υποστεί ε, κατατρεχμό. Δυστυχώς πάλι τα αρνητικά παραδείγματα μου έρχονται πρώτα στο νου, αλλά είναι αναπόφευκτο το τι συμβαίνει στο Αζερβαϊτζάν με τις αντιφρονούντες, με τους ακτιβιστές στην Λευκορωσία, με τη δίωξη δημοσιογράφων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Ουκρανία. Πριν από τρεις μέρες, μια γυναίκα που εργάζεται σε ανθρωπιστική οργάνωση απήχθη στο Λουγκάνσκ από τις ένοπλες ομάδες εκεί. Κατηγορήθηκε ότι είναι κατάσκοπος Εργάζεται για την Μέρση Κόρψη, είπανε, αλλά είναι Ουκρανοί ε, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική οργάνωση. Παράλληλα, μιλώντας για την Ουκρανία, Η άλλη όψη της έναπλης σύγκρουσης είναι ότι μία από τις τρεις γυναίκες δημάρχους πόλεων της Ουκρανίας πριν τον πόλεμο, η Νιέλε Στέπα, μετετράπησε από διοπιμπαίο τράγο. Είναι σε κράτηση εδώ και 1,5 χρόνο. Κατηγορείται ότι υποστήριξε τα φιλορωσικά αισθήματα και το τα υποδάβλιζε. Δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα, πραγματικές αποδείξεις για να αποδειχθεί αυτή τη δράση Πέρα από το ότι ήταν γυναίκα δήμαρχος της, Τάν, της πόλης του Σλαβιάνσκ στην ε, Ανατολική Ουκρανία. Θετικά παραδείγματα μόνο από την κοινωνία των πολιτών έχουμε. Διότι παρά τις αντικσότητες, παρά τις διώξεις, παρά τις απειλές σε πολλές από αυτές τις χώρες, εκεί οι ομάδες των γυναικών οργανώνονται. Στην Ουκρανία λόγου χάρη. Εγώ ήμουν στον Πετρόφσκ τους τελευταίους 6 μήνες Είχα γυναίκες εσωτερικά μετατοπισμένες ε, που είχαν ε, ε, καταφέρει να επιβιώνουν πολύ λίγα. Οι οποίες είχαν φύγει από το Λουγκάνσκ για να σώσουν τις ζωές τους. Οι οποίες είχαν καταφέρει να οργανωθούν σε αυτές τις μικρές οργανώσεις, τις ε, μικρές ομάδες εσωτερικών μετατοπισμένων όχι μόνο γυναικών, όλων όσων έχουν πληγεί από τη σύγκρουση και εμείς από την διεθνή κοινότητα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το δίχτυ διεθνούς προστασίας με ένα φόρουμ, με συναντήσεις συντονισμού ε, για την Ουκρανία, εντός της Ουκρανίας, προσπαθώντας να εμπλέξουμε αυτές τις αυθορμήτως οργανωμένες γυναίκες από τις οργανώσεις των εσωτερικών μετατοπισμένων. Λειτουργήσαν κάπως σαν βαρόμετρο με μία φωνή πραγματικά ε, σημαντική ε, για να δούμε τι κάνουν οι χώρες μας και αν ε, έχουμε τις σωστές επιδιώξεις με τις ανθρωπιστικές μας κινήσεις, τις βοήθειες, με τη χρηματοδότησή μας και τις σχετικές πρωτοβουλίες πετυχαίνουμε αυτά που χρειάζονται. Αυτό μπορούσαμε να δούμε χάρη σε αυτές. Η ψήφος μου λοιπόν πηγαίνει στην κοινωνία των πολιτών και τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Οι δύο ερωτήσεις ήταν ποιοι οι λόγοι για να είναι τόσο ισχυρά και δημοφιλή αυτά τα κινήματα που είναι συντηρητικά και κατά των δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Η βασική μου εξήγηση είναι ότι τα κινήματα αυτά δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το φύλλο. Βεβαίω επιτίθενται στι πολιτικέ ισότητα των φύλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιπτώσει για την ποιότητα τη ισότητα των φύλων και για τι γυναίκε. Έχουν τεράστιε συνέπειε σε όλη την Ευρώπη. Όμω δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Περισσότερα αφορούν τη δημιουργία μιας νέας θεώρησης για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να φασίζεται σε διαφορετικέ αξίε από αυτέ που τώρα υπερασπιζόταν η πυρό μα. Ο τρόπο που το βλέπω, η... το γεγονό ότι είναι τόσο δημοφιλή τα κινήματα αυτά, ε, προκύπτει από την ανασφάλεια. Οι άνθρωποι έχουν ανασφάλειε, φοβούνται την ε, παγκοσμιοποίηση, οι ανισότητε. η εντύπωσή τους ότι δεν έχουν αρκετή, ότι αντιμετώπιση με αρκετή αξιοπρέπεια, δεν γίνεται σεβαστή αξιοπρέπειά τους και ότι έχουν πάρει απόσταση από τις πολιτικές ελίτ. Είναι τόσο ισχυρά τα κινήματα αυτά γιατί παριστάνουν ότι δίνουν τις σωστές απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Λένε εντάξει, αισθάνεστε ασφαλείς. Εμεί θα σα δώσουμε ασφάλεια με μια παραδοσιακή οικογένεια. Ή η παγκοσμιοποίηση αισθάνεστε, αισθάνεστε ότι σα απειλεί. Πώ αισθάνεστε με την αλληλοδιασύνδεση με άλλε χώρε. Δεν σα αρέσει να πάμε πίσω στην εθνική μα κοινότητα γιατί θα ξαναβρείτε την ασφάλειά σα. Ή σα φοβίζουν οι γρήγορε πολιτιστικέ αλλαγέ. Να πάμε πίσω στου παραδοσιακού ρόλου των φίλων, α πούμε, και ότι το καθεξή. Η σα φοβιζουν οι γρηγορε πολιτιστικε αλλαγε να παμε πισω στου παραδοσιακου ρολου των φιλων α πουμε και ουτω καθεξη η απαντηση μου λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα για το τι μπορεί να γίνει είναι Ίσως να θέλετε κάτι πιο ακριβές, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε και να επεξεργαζόμαστε αυτά τα αντιεπιχειρήματα όπως είπατε. Να βρούμε κάτι να λέμε που να έχει να κάνει με την πολιτική διάσταση του θέματος. Πολιτικές και μέσα για τα δικαιώματα των γυναικών δεν αρκούν τώρα Έχουμε φτάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο στην ιστορία που τα κινήματα αυτά επιτίθενται και αμφισβητούν αυτές τις ίδιες τις πολιτικές. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να ε, αντιμετωπίσει την αντίσταση σε αυτές τις πολιτικές απλώς εφαρμόζοντας τις πολιτικές. να πάει παραπέρα. Η δική μου λοιπόν πρόταση θα ήταν να δώσουμε καλύτερες απαντήσεις σε αυτές τις απειλές. Έλλειψη ασφάλειας, ανισότητες, παγκοσμιοποίηση καλύτερες αποκρίσεις σε αυτές τις απειλές από τους νέους συντηρητικού και τους φονταμεταλιστές, τους θρησκόληπτους. Είναι δύσκολο να σας ε, ξεχωρίσω μία και μόνη πρακτική, αλλά αυτή που σίγουρα θα συνέστηνα είναι τα κινήματα της βάσης να τα προβάλλουμε όσο το δυνατό περισσότερο, διότι καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τις απειλές που έχουν να αντιμετωπίσουν, τις αισθάνονται και τις ζουν στην καθημερινότητα. Εκείνοι καταλαβαίνουν να μιλάμε σωστά για την ισότητα, αν χειριζόμαστε όλα αυτά τα θέματα σωστά και να υπάρχει απήχηση και στο κοινό. Βεβαίω, πρακτικά η απάντησή μου δεν είναι πολύ απλό να χρησιμοποιηθεί. Στρατηγικά δεν είναι εύκολο αλλά τα κινήματα αυτά μόλις τώρα αρχίσαμε να τα μελετάμε και είναι ίσως μία αρχή. Ε, Ευχαριστώ. Να επανέλθω σε τρία ερωτήματα που τέθηκαν. Καταρχάς αναφέρεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τιμωριό. Οι ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, ε, ανθρώπινα δικαιώματα ως αντάλλαγμα για το εμπόριο, το 2011 ε, είχαμε μία ανακοίνωση και άλλη μία τον περασμένο Νοέμβριο. Αν τη συγκρίνουμε θα δούμε ότι υπάρχει μία αλλαγή. Έχουμε περάσει από τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σταθεροποίηση, την ε, φάταξη της τρομοκρατίας ε, και την ασφάλεια. Έχει αλλάξει η οπτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά χρησιμοποιεί τη δύναμή της για να αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο όταν διαπραγματεύεται από κοινού συμφωνημένες προτεραιότητες εταιρική σχέσης. Η διοκτησία λοιπόν εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιβάλλει κάτι μέσα στα πλαίσια του ΙΕΠ. Είναι μια κοινή πλατφόρμα για να ε, συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε εμπορικές συμφωνίες. Αυτή λοιπόν η πλευρά του ΙΕΠ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας δεν θα εξαφανιστεί παραμένει για κάποιες χώρες όπου είναι δυνατόν, την Ισία, η Ορδανία. Ε, το είδατε εκεί, στην ε, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, αλλά δεν είναι παρούσα σε περιπτώσεις όπως της Αιγύπτου. Για την κοινοβουλευτική διπλωματία επίσης, να πω ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ε, όπως θέλουμε, να έχουμε συναντήσεις κοινοβουλευτικές και να πηγαίνουμε και στο πεδίο ε, όχι για να ε, συναντήσουμε μόνο συναδέλφους, ε, για να δούμε την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου και να δούμε και τη σύνδεσή του με τον πραγματικό κόσμο, γιατί πολλές φορές γίνονται εκλογές εντός εισαγωγικών. Δεν πρέπει να διστάζουμε να προκαλούμε και τις αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης που υπάρχουν για την κάθε χώρα χωριστά. Για τις βέλτιστες πρακτικές Τέλος, να πω ότι πρόσφατα πήγα στην Ιορδανία για μια ε, περιφερειακή συνάντηση. Έγινε μια παρουσίαση του σχεδίου δράσης για το φύλλο του ΓΚΑΠ στην Ιορδανία. Ήταν πολύ ολοκληρωμένη και πολλά υποσχόμενη. Όμως, να πω ότι υπάρχουν δύο κίνδυνοι που πρέπει να αποφύγουμε να ε, έχουμε δηλαδή μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο εστίασης και να το ξεχνάμε μόλις το αποφασίζουμε και μετά να, να αποφύγουμε απλώς να τσεκάρουμε κουτάκια ότι αυτό είναι το σχέδιο δράσης, ε, τσεκάραμε όλα τα κουτάκια ότι τα κάναμε και ας πάμε στην πραγματική δουλειά. Αυτή είναι η δύο κίνδυνοι που βλέπω στην εφαρμογή. Και αυτό ξέχασα να το πω στην παρουσίασή μου. Αυτό, το προτείναμε, αυτό που προτείναμε ήταν η επικεφαλής των αντιπροσωπιών να είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή. Βέβαια, ε, όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο ότι όταν οι ηγέτες θα αναλαμβάνουν τα ενία θα λαμβάνουν τα σοβαρά υπόψη εφαρμογή το πρόβλημα με τον ΚΑΠ ήταν ακριβώς ότι τα υψηλότερα, οι υψηλότερες βαθμίδες ε, των αντιπροσωπιών της Κοσμισιόν ε, και των ε, λοιπόν εμπλεκόμενων δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους το θέμα. Θα ξεκινήσω απαντώντας σε αυτό που είπατε, ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών θα λογοδοτούν για, αυτό, για αυτή την εφαρμογή. Έχει να κάνει με την εξωτερική δράση έχει καλυφθεί βέβαια από εσά το θέμα. Τώρα για τα άλλα ερωτήματα σχετικά με τις συμφωνίες εμπορίου και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επανέλθω γραπτός γιατί περιλαμβάνει και τη Γενική Διεύθυνση Trade. Είναι δύσκολο λοιπόν να απαντήσω εκ μέρους και άλλων διευθύνσεων. Για το θέμα του ρόλου των γυναικών στην Παλαιστίνη υπάρχουν διάφορα project που έχουν υποστηριχθεί, αλλά και αυτό θα σας το δώσω γραπτός για να έχετε μια πλήρη απάντηση. Τρίτο ερώτημα σχετικά με το αν μπορούμε να έχουμε μία βέλτιστη πρακτική που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Είναι καλό να έχουμε καλές πρακτικές και να μαθαίνουμε από αυτές, αλλά όταν μιλάμε για την ισότητα των φύλων πάντοτε πρέπει να κοιτάμε το συγκείμενο, το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν χρειάζεται απλώς να κάνουμε copy-paste, γιατί πολλές φορές αυτό είναι λάθος και βιώνουμε μια ματέωση. Ε, προσπαθούμε κάτι πετυχημένο να το επαναλάβουμε αλλού και δεν γίνεται. Επίσης, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς τις προσδοκίες μας. Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα τέτοιο σχέδιο δράσης μέσα σε πέντε χρόνια με τα θέματα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι. Ένα άλλο θέμα που πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με άλλους, λοιπόν. Για το θέμα της μετανάστευσης, ε, να συνταχθώ με τους συναδέλφους και να πω ότι θα επανέλθω και για αυτό το θέμα γραπτός, αν μου επιτρέπετε, για την εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό θέμα. Περιλαμβάνεται και στο σχέδιο δράσης για το φύλλο, αλλά και στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων. Ειδικά όταν μιλάμε για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, όπου η παράδοση, η εκπαιδευτική είναι λίγο διαφορετική από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ε, αυτή η περίοδος η κομμουνιστική που όλοι είχαν ε, εκπαίδευση, αλλά ξεχνάμε ε, εξαιρέσεις όπως τους Ρωμά κτλ. Ε, καλό είναι λοιπόν να προωθούμε την ισότητα των φύλων και μέσα από αυτά μέσα από αυτές τις δράσεις για την εκπαίδευση μπορεί να προωθούμε ακόμα περισσότερο το θέμα της ισότητας των φύλων. Σας ευχαριστώ λοιπόν που το αναφέρατε. Είναι κάτι που έχει μπει ε, σε επεξεργασία και θα το χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους μας για τις πολύ μεστές ε, και άρτιες παρουσιάσεις που μας έκαναν. Τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να αντλήσω κάποια συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου το συμπέρασμα μπορεί να συνοψιστεί στο εξή. Τι συμπέρασμα, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι να ολοκληρώσουμε αυτό το ζήτημα. Πόρο απέχουμε από την επίλυση αυτού του θέματο και θα πρέπει να δίνουμε τι προσπάθειές μα για περισσότερη στήριξη, περισσότερη συνεργασία, περισσότερη συνδρομή. Εντοπίσαμε κάποιου βασικού ε, κέριου τομεί. Επιμείναμε πολύ στην ανάγκη τη παρουσίας των γυναικών σε θέσει ε, ε, υψηλόβαθμε λήψη αποφάσεων και όπω είπε και η κυρία Κατσάροβα θα πρέπει να έχουμε συνεργασία σε εθνικό επίπεδο από το τοπικό μέχρι το κυβερνητικό, να τονίσουμε και την ανάγκη της εξωτερικής πολιτικής, να αναδείξουμε και να εξάρουμε το ρόλο των γυναικών όχι μόνο για την επίλυση των διαφορών, για την πρόληψη ε, των σειράξεων, αλλά και για την εξασφάλιση ε, μιας πιο βιώσιμης ειρήνης ε, και την εγγύηση της ασφάλειας. Είναι, σημαντικά για, είναι σημαντικός για όλα αυτά ο ρόλος και η παρουσία των γυναικών. Επίσης υπάρχουν στη βάση κάποια κινήματα που φαίνεται ότι βρίσκονται σε έξαρση και προσπαθούν να αμφισβητήσουν αυτό το ρόλο των γυναικών ε, συνδέοντας την επαναφορά σε παραδοσιακές φαλοκρατούμενες απόψεις με το θέμα της ανασφάλειας και του φόβου. Επίσης μιλήσατε για το θέμα των βέλτιστων πρακτικών, τη θέση της κοινωνίας των πολιτών, των μικρών ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων που καθημερινά δίνουν μάχη για να προσπίσουν τη θέση των γυναικών. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη και τη δική τους συνεισφορά. Επίσης, συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, γυναική επιχειρηματικότητα. Έχουμε το πρόγραμμα «Γυναίκες στις επιχειρήσεις», «Women in Business». Επίσης, βασικό θέμα της ειρήνης, ε, για την εδραίωση της ειρήνης ή βία κατά των γυναικών. Πολύ θετική η ομιλία του κυρίου Φόρες, γιατί ξεκινήσαμε από θετικά παραδείγματα και θέσαμε κάποιες πιο γενικέ ερωτήσεις που μας ε, ενδιαφέρουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, εγώ αναφέρθηκα στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά υπάρχουν και άλλες του ΩΣΑ, για παράδειγμα. Πολύ δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με μονομένα τα κράτη-μέλη. Και φυσικά δεν ξεχάσαμε και το ζήτημα της μετανάστευσης και την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Πολύ σημαντικό και το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να γενικεύουμε, να αποφύγουμε τις γενικεύσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδιαιτερότητες και στα διαφορετικά πλαίσια. Το πρωταρχικό πάντως μήνυμα είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη, πολύ έργο, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να τις εντείνουμε και να τις βελτιώσουμε, θα έλεγα εγώ. Όχι απλώς να τις εντείνουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Πολύ χρήσιμες, πολύ σημαντικές οι, οι, οι απόψεις, οι προτάσεις για την θέση των γυναικών στην πολιτική γειτονία προς Ανατολάς και προς τον Νότο και τις την Ανατολική και Νότια Εταιρική Σχέση. Και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με τους και συζητητές και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής των Γυναικών. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν είχαμε προβλέψει αρχικά ότι θα παρατείναμε τόσο πολύ τη δημόσια κρόση. Σας ευχαριστώ πάντως και σήμερα για τη συμβολή σας. Καλό σας απόγευμα.